Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα έντυπο στην, ε, από την μερίσια διάταξη που είχε λάθος αίθουσα απάνω και ίσως γι' αυτό να μην έχουν έρθει οι διάφοροι. ο κύριο Μάντες που είναι υπεύθυνο για τη μελέτη της ε, Κομισιόν Λύπη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αφού έρθει. Θα φροντίσω να τον πάρω με το κινητό μου, να έρθει. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ ήδη. Και η κυρία Κέπαρτ και εγώ είμαστε εδώ. Βέβαια στον αντίποδα ο ένας από τον άλλον, σε αυτή την αίθουσα. Τι να κάνουμε, αλλά περιμένουμε λίγο. Θα πρέπει να περιμένουμε και αυτό λόγω της αλλαγής ε, αίθουσας που έχουμε κάθε τόσο λόγω των ακροάσεων κλπ. Uh, Καλημέρα και πάλι. Έχουμε εδώ τον ε, κύριο Μάντες που είναι και συγητή μας ε, για το θέμα της επισήμας κλωστοφατουργικών προϊόντων. Και η κυρία Κέμπαρτ είναι εδώ που εκπροσωπεί την κυρία Σαλτεμόζη, η κυρία Ρούλη είναι εδώ επίσης και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Δεν ξέρω αν κυρία Μακλάκ είναι εδώ. Όχι. ο κύριος Σαβίνη είναι εδώ όμως, ανταυτού. Συνεπώς, το πρώτο θέμα που έχουμε σήμερα το πρωί είναι μια παρουσίαση, μια μελέτη της Επιτροπής για την ε, επισήμανση κλωστιφαντουργικών προϊόντων. Υπάρχει εδώ, έχουμε ένα αντίγραφο και η κυρία Μπενίτα Κίτσπιτς είναι εδώ για να παρουσιάσει εκ μέρου του Rambo Consulting την, ε, τα συμπεράσματά τους και ίσως να απαντήσει και σε ερωτήσεις. Οπότε σας δίνω το λόγο, θα χρησιμοποιήσετε και διαφάνειες, έτσι, παρακαλώ. Η ε, κυρία Γκέπαρθ πρώτα όμως. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω. Οι διερμηνείς μόλις μου είπαν ότι δεν έχουν έγγραφα και είναι σημαντικό να έχουν και αυτή την παρουσίαση. Και εγώ στη δική μου θέση, ούτε κι εγώ βρήκα στη θέση μου τα σχετικά έγγραφα. Δεν ξέρω, ίσως τα slides να πρέπει να τα δώσετε ή θα μας βοηθήσουν οι διαφάνειες για να παρακολουθήσουμε. Περιμένουμε τις ε, διαφάνειες σου. Ωραία. Η κυρία Μακλάρκιν είναι εδώ, που είναι επίσης σκιώδης ηγήτρια για την ομάδα ICR, για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή μοιράζουμε αντίγραφα των διαφανειών που θα λάβουν και οι διερμηνείς. Προτείνω να ξεκινήσετε. Εάν όλοι οι βουλευτές έχουν λάβει τα αντίγραφα, μπορείς να ξεκινήσεις και να περιμένεις να βάλουμε πρόσκληση την τεχνολογία. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Καλημέρα όπως ε, αναφέρθηκε, ανατέθηκε στην Κομισιόν να εξετάσει ε, τις ε, συνέπειες που έχουν να κάνουν με την επισήμανση των γλωσσοφαντουργικών προϊόντων. Εκπονήσαμε μία μελέτη αντικτύπου σε περίπτωση εισαγωγής των μέτρων που προτείνουμε και εξετάστηκαν οι θετικές και αρνητικές πτυχές. Οι απαιτήσει ως προς την επισήμανση ε, έχουν να κάνουν με την ε, μεταχείριση του προϊόντος, ε, την χημική σύσταση, την προέλευση, την, οικολογική, την περιβαλλοντική επισήμανση κλπ. Έχουμε μια πρόσφατη, ένα πρόσφατο κανονισμό για την κλωστοφατουργία που υιοθετήθηκε ε, τον Ιανουάριο του 2009 από την ε, Επιτροπή εξετάστηκαν και άλλες ε, δυνατότητες. Δεν ήταν λοιπόν στόχος μας να αλλάξουμε την προηγούμενη πρόταση, αλλά να βρούμε ένα μηχανισμό που να παρέχει πιο πλήρη ενημέρωση στον καταναλωτή. Η χρησιμότητα της πρότασης αυτής Ε, στόχο έχει να αποτελέσει βάση για μελλοντικέ ε, νομοθετικές προτάσεις. Γενικά βρήκαμε ότι οι ενώσεις καταναλωτών γενικά δεν ε, παρακολουθούν στενά την επισήμανση κλωστοφατουρικών προϊόντων με εξαίρεση την χημική σύσταση. Ο λόγος ο λόγος γι αυτό είναι ότι δεν θεωρείται ότι η κακή επισήμανση, ε, με εξαίρεση την χημική σύσταση, ε, μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Γενικά, ε, ο βιομηχανικός τομέας ήταν υπέρ προαιρετικού συστήματος. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι θεωρεί ότι τα υποχρεωτικά συστήματα συνεπάγονται και σημαντικό κόστος αναφερθώ λεπτομερώς στο ποιο θα είναι το κόστος και για τα κράτη-μέλη ήταν σαφές ότι τα υποχρεωτικά συστήματα θα αυξήσουν τις απαιτήσει για επιτήρηση της αγοράς και κάναμε μια ε, σχετική μελέτη και διαπιστώσαμε ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν ε, πρόβλημα όσον αφορά την, την τήρηση των ε, υποχρεώσεών τους ε, στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους. Ε, οι αρχές επιτήρησης της αγοράς λοιπόν δεν θα συναντήσουν δυσκολίες στην περίπτωση αυτή. Όσον αφορά την επισήμανση για τη φροντίδα του προϊόντος, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα δύο τρίτα έχουν προαιρετικά συστήματα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που περιλαμβάνουν ε, και ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, έχουν υποχρεωτικά συστήματα σύμφωνα με το ISO 3758, το οποίο σημαίνει ότι λίγο πολύ το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Η ενός καταναλωτών είναι υπέρ εναρμονισμένου καθεστώτος, διότι έτσι οι καταναλωτές θα ε, συναντούν τα ίδια σύμβολα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, έτσι θα γνωρίζουν τον τρόπο σωστής φροντίδας του προϊόντος. Το υποχρεωτικό σύστημα βρήκε επίσης υποστήριξη και ο βασικός λόγος είναι ότι με προαιρετικό σύστημα οι εταιρείε μπορούν να αποφασίσουν εάν θα το εφαρμόζουν ή όχι το οποίο σημαίνει ότι η βεβαιότητα του καταναλωτή δεν είναι τόσο, τόσο υψηλή όσο είναι ε, με ένα υποχρεωτικό σύστημα. Ε, ο βιομηχανικός τομέας και οι φορείς τυποποίησης ε, είναι κατά ενός υποχρεωτικού καθεστώτος, διότι θεωρούν ότι το παρόν καθεστώς λειτουργεί μια χαρά και λόγω του επιπλέον κόστους που θα συνεπάγεται ένα υποχρεωτικό σύστημα. Ε, οι δαπάνες αυτές συνδέονται κυρίως με ε, πρόσθετες δοκιμές. Η Κομισιόν θεωρεί ότι αν η επισήμανση για τη φροντίδα του προϊόντος γίνει υποχρεωτική, τότε Οι λιανοπολιτέ θα πρέπει να κάνουν περισσότερους ελέγχους από αυτούς που ήδη κάνουν, διότι ε, θα θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Το κόστος γενικά το φέρνουν οι καταναλωτές σε περίπτωση επιπλέον επισήμανσης. Εάν ε, μία ή να μπορεί να πληθεί στους 30 βαθμούς αλλά η ε, βιομηχανία ε, θέλει να είναι πιο επιφυλακτική και γράφει ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε στεγνό καθάρισμα, αυτό συνεπάγεται πλέον κόστος για τον καταναλωτή. Επίσης υπάρχουν κάποιες νομικές συνέπειες και η βασική νομική συνέπεια του υποχρεωτικού συστήματος συνδέεται με το γεγονός ότι ε, τα σύμβολα αυτά είναι αντικείμενο, αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Genotext ε, και ε, αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλη την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι για να συμμορφωθούν με την ομοθεσία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρώνουν την Genotex για να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ένα σύστημα που έχει να κάνει με κατατεθέντα σήματα τα οποίο θα πρέπει να λυθεί σε περίπτωση που η επισήμανση για τη φροντίδα γίνει υποχρεωτική. Ε, το πιο σημαντικό θέμα για τις ε, ενός καταναλωτών είναι ε, η χημική σύσταση, διότι θεωρούν ότι το θέμα των ε, χημικών ουσιών στα υφάσματα δεν καλύπτεται επαρκώς από την οδηγία REACH. Δεν καλύπτονται όλες τι τεχνολογίες και υπάρχουν ακόμα πολύ ψηλά ποσοστά κάποιων χημικών ουσιών σε κάποια υφάσματα. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα νομοθεσίας, υπάρχει και ένα πρόβλημα συμμόρφωσης με την νομοθεσία. Οι ενώσεις καταναλωτών επίσης επισήμαναν ότι η επισήμανση δεν αρκεί, μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί για να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με το τι περιέχεται σε ένα προϊόν και οι ενώσεις καταναλωτών πιστεύουν ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ο καταναλωτής όμως δεν θα πρέπει να βασίζει την απόφαση του στην επισήμανση διότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό έναν κίνδυνο για την υγεία του και δεν θεωρεί δεν θεωρούν οι ενώσει καταναλωτών ότι είναι ε, ε, ευθύνη του καταναλωτή αυτό να λάβει τι αποφάσει αυτέ με βάση την ε, επισήμανση. Η επισήμανση δηλαδή αποτελεί βοήθεια, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί στη βάση για τι αποφάσει του καταναλωτή. Υπάρχει και το θέμα τη συμμόρφωση. Οι αρχέ εποπτεία τη αγορά θα πρέπει να ελέγχουν τα προϊόντα. Όσον αφορά το κόστο για τη βιομηχανία, σε περίπτωση που σε περίπτωση υποχρεωτική σήμανση ε, των χημικών ουσιών ε, θα συνδέεται με ε, πρόσθετε δοκιμέ για τι ουσίε αυτέ. Αυτή τη στιγμή γίνονται δειγματοληπτικέ δοκιμέ, αλλά σε περίπτωση εισαγωγή ενό συστήματο επισήμανση θα πρέπει να γίνονται πιο πλήρεις δοκιμέ. Η βιομηχανία δεν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα επιφέρει προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή. διότι όλοι οι υπεύθυνοι παραγωγοί ούτως ή άλλως ε, συμμορφώνονται με την νομοθεσία, ενώ αυτοί που ενώ οι ανεύθυνοι δεν ε, διστάζουν να βάλουν λάθος πληροφορίες σε μια ετικέτα προϊόντος. Επίσης ε, φοβούνται ότι εάν αναφέρουν σε μια ετικέτα ότι ε, το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει κάποιες χημικές ουσίες, ο καταναλωτής δεν θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Όσον αφορά την ηλεκτρονική επισήμανση που έχει να κάνει με την με το ηλεκτρονικό σώσιμο πληροφοριών πάνω σε ένα ε, ένδυμα ε, έχει να κάνει με την διαχείριση της ε, τροφοδοτική αλυσίδας. Φαίνεται ότι ε, απαιτείται περαιτέρω τεχνολογική πρόοδος για να μειωθεί το, η τιμή, το κόστος των ετικετών αυτών. Το κόστος εισαγωγής του τσίπ είναι χαμηλό, αλλά αλλά συνδέεται με κάποια επιπλέον συνδέεται με κάποιο επιπλέον κόστος. το βασικό πρόβλημα για τους καταναλωτές είναι ε, ο σεβασμός ιδιωτικής ζωής. Οι ενώσεις ε, καταναλωτών ε, πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς τον καταναλωτή και να του γίνονται διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες αγορές του λόγω του τσιπ. Όσον αφορά την ε, επισήμανση σε πολλές γλώσσες. Ε, φαίνεται ότι το παρόν καθεστώς ε, μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές. Οι ενώσεις καταναλωτών θα προτιμούσαν υποχρεωτική ε, πολύγλωση επισήμανση για όλες τις ετικέτες, αλλά αναγνωρίζουν ότι γενικά οι καταναλωτές δεν επηρεάζονται πολύ από το παρόν σύστημα, η βιομηχανία είναι ικανοποιημένη από το παρόν σύστημα. Η παρούσα στρατηγική είναι να παρέχονται πληροφορίες στην γλώσσα των αγορών στις οποίες στοχεύουν οι επιχειρήσεις. Και ε, υπάρχει ε, βέβαια το θέμα της αλλαγής ετικέτας ε, όσον αφορά τη χώρα προέλευσης και αυτό εξετάστηκε και αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς συζήτησης το 2005 υποβλήθηκε σχετική πρόταση της Επιτροπής που δεν έχει περάσει ακόμα από το Συμβούλιο όμως. Το όφελος για τους καταναλωτές όσον αφορά την επισήμανση χώρας προέλευσης περιορίζεται στην καλύτερη ενημέρωση, διότι δεν ε, συνεπάγεται κίνδυνο για τους καταναλωτές σε περίπτωση λάθους επισήμανσης. Αλλά, για παράδειγμα, ένα πουκάμισο μεγάλο μέρο ενό ποκαμίσου μπορεί να, ε, ε, κατασκευαστεί στην Κίνα και τελικά η τελική ραφή να γίνει σε άλλη χώρα ε, και αυτό να μην μπορεί να καλυφθεί με τον παρόντα ορισμό της επισήμανσης της χώρας προέλευση. Ε, με την επισήμαση της χώρας προέλευσης υπάρχει ίσως οριακά ένα πλεονέκτημα για τα, τους παραγωγούς εντός των κρατών μελών, διότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα ε, ευρωπαϊκής προέλευσης, διότι ε, θεωρούνται καλύτερης ποιότητας. Αλλά ε, τα, η βιομηχανία είναι διχασμένη στο θέμα αυτό και μεταξύ των κρατών μελών και εντός των κρατών μελών και φαίνεται ότι τελικά διαφέρει η, διαφέρουν οι απόψει των μεμονωμένων εταιριών μεταξύ τους. Η τεκμηρίωση και ο εκτελονισμός ε, επιφέρουν ε, επιπλέον ε, δαπάνες που μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα των εισαγωγέων και ε, ε, αυτομάτως γίνεται μετακύληση στον καταναλωτή των δαπανών αυτών. Όσον αφορά την οικολογική επισήμανση, οι ενώσει καταναλωτών πιστεύουν ότι οι καταναλωτέ ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον τομέα αυτών και ένα όφελο για του ε, καταναλωτέ είναι ότι το ε, ένδυμα είναι απαλλαγμένο από χημικά και ότι συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντο αγοράζοντα τέτοια προϊόντα. Ωστόσο, το κόστο ε, για μια οικολογική επισήμανση είναι σημαντικό. Πρέπει να πληρωθούν τέλη, πρέπει να γίνουν χημικέ δοκιμέ και πρέπει να γίνονται και επιθεωρήσει ώστε να διαπιστώνουν διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις πράγματι ε, συμμορφώνονται με τις απαιτήσει για επισήμανση. Από την πλευρά λοιπόν της βιομηχανίας ε, οι ε, καταναλωτές θα πρέπει να ενδιαφερθούν περισσότερο για το θέμα αυτό προτού η βιομηχανία να αρχίσει να επενδύει στον τομέα αυτό. Ο τελευταίος τομέας που εξετάσαμε ήταν η επισήμανση που έχει να κάνει με τα μεγέθη. Ο εναρμονισμός συστήματος μεγεθών έχει καλυφθεί με έχει καλυφθεί με ένα σύστημα προαιρετικό που λέγεται EN13402. Ε, είναι προαιρετικό όμως, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα διαφορές όσον αφορά τα μεγέθη. Ε, από πλευρά των καταναλωτών ε, δεν είναι πολύ ανησυχητικό το ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα καθορισμού του μεγέθους. Είναι κοινή πρακτική ο καταναλωτής να ρωτάει στο κατάστημα τι μέγεθος να ε, αγοράσει, τι μέγεθο του κάνει. Ε, αλλά βέβαια οι καταναλωτέ όταν του ρωτήσαμε είπαν ότι θα θέλανε ένα εναρμοσμένο σύστημα διότι αυτό θα διευκολύνει τη ζωή τους. Ε, θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα που να αποτελεί αντικείμενο συνένεση διότι αλλιώς θα μπορούσε να είναι πρόβλημα το ποιο σύστημα θα επιλεγεί. Οι περισσότεροι ήταν υπέρ ενός τέτοιου συστήματος παρά το υψηλό κόστος που θεώρησαν ότι θα επιφέρει κάτι τέτοιο. Ούτω ή άλλω μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο όπου θα χρησιμοποιούνται παράλληλα δύο συστήματα και θα πρέπει επίση να υπάρξει κάποια εκστρατεία για να γνωρίσουν οι καταναλωτέ το νέο σύστημα. Να συνοψίσω σύντομα. Η χημική επισήμανση, όπως σας ανέφερα, είναι ε, το το πιο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να εξεταστεί τουλάχιστον από πλευράς των καταναλωτών. Η υγεία του καταναλωτή διακυβεύεται, ενώ οι άλλοι τομείς μπορεί να προκαλούν κάποια ενόχληση στους καταναλωτές εάν δεν είναι εναρμονισμένοι, αλλά δεν φαίνεται να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Χθε το απόγευμα η Επιτροπή είχε βιντεοδιάσκεψη διαρκεία μια ώρα με το Παρίσι, με ταυτόχρονη διαρμηνία και εικόνα. Τέλεια κάλυψε τι υπηρεσίε. Πώ δεν μα συνδέσουν έναν υπολογιστή για να έχουμε προβολή διαφανιών, οι ίδιοι τεχνίτε, η τεχνική δεν ξέρω πώ γίνεται. Χρειάζεται κατάρτιση. Για τι επόμενε δύο παρα... παρουσιάσει, α είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τι διαφάνειε. Είχαμε τι διαφάνειέ σα δεν αναφερθήκατε στον οργανισμό σας. Και δεν βρήκα τίποτα στη μελέτη. Ε, να μας πείτε ποιοι είστε. Δεν παρουσιάσατε τον φορέα που εκπροσωπείτε. Ναι, βεβαίω. Rumble Management Consultant. Είναι συμβουλευτική εταιρεία. Κάνει αξιολογήσεις και μελέτες. Κυρίως για δημόσιους φορείς. Κάνουμε πολλή δουλειά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Ευρωκοινοβούλιο και για εθνικούς δημόσιους φορείς στη Δανία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Σουηδία και την Ορβηγία. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στον αφορά τις αξιολογήσεις, τις μελέτες και τις μελέτες ε, συνεπιών και αντιχτύπου. Πρόεδρος. Θα έπρεπε να έχετε ένα σημείωμα για τους ε, αναδόχους που αναλαμβάνουν τις μελέτες. Έχουμε τους εισηγητές και τους χιώδεις εισηγητές που ασχολούνται με το θέμα. Ας γίνει ένας γύρος ερωτήσεων. Έχουμε στις 10 το δεύτερη παρουσίαση, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά θα σημειώσουν ε, οι σύμβουλοι τις ερωτήσεις σας. Χουάν Μάντες που είναι αριστερά, που είναι συγητής για την πρόταση, ίσως ε, θα μπορούσε να προβεί σε ένα-δύο σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για τη μελέτη. Δεν είναι λεπτομερής η μελέτη ακόμα, αλλά είναι αδύνατο τόσο σύντομα να γίνει κάτι τέτοιο. Δείχνει την κατεύθυνση δείχνει τι θέλουν οι καταναλωτές, τι θέλει η βιομηχανία. Και αυτές οι πληροφορίες μας αρκούν για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Δύο. Πολλές βεβαίως, αλλά δύο βασικά. Οι εικόνες του Ginatex για να πώς προσέχει κανείς το ένδυμα Αυτά τα εικονίδια είναι τα πιο γνωστά. Αναφερθήκατε σε θέματα πνευματικών, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, κόστος, που η Gina ζητά χρήματα, δικαιώματα. Εξετάσατε ποιε είναι οι δαπάνε. Θα είναι πιο ψηλέ από ό,τι τώρα. Διότι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια Ginatex στα κράτη-μέλη σε αβιομηχανία πρέπει να πληρώσετε δικαιώματα στη Τέξ και σε κάποιον εθνικό φορέα. Υπάρχει διαφορά σε κόστος αν εισαγάγει αυτό το σύστημα βιομηχανία. Πρώτο ερώτημα ήταν αυτό. Δεύτερο. Ετικετοθεσία για το μέγεθος. Δεν θεωρείται πρόβλημα σε εθνική βάση από τον καταναλωτή. Αλλά στις πωλήσει μέσω διαδικτύου θα μπορούσε να είναι πρόβλημα αυτό. Μιλήσαμε με την Κούτσι στο Μιλάνο και θέλανε να υπάρχει ένα μέγεθος για την Ευρώπη. Είπαν παράγουμε την ιστορική αγορά. Και δεν είναι απλό για μας να προσθέτουμε όλα αυτά τα διαφορετικά μεγέθη για κάθε χώρα στο ίδιο ένδυμα. Εμείς παράγουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι πλέον για πολίτες ξεχωριστών χωρών. Είπατε ότι χρειάζεται χρόνος. Χρόνος για να επανεκπαιδευτεί και η βιομηχανία και οι καταναλωτές. Μπορείτε να πείτε πόσο χρόνος προβλέπετε ότι χρειάζεται. Διότι αν θέλουμε να έχουμε ένα πρότυπο ευρωπαϊκό για τα μεγέθη, για τα ρούχα και για τα παπούτσια, θα χρειάζεται μεταβατική περίοδος. Για να προσαρμοστεί ο κόσμος στην ετικέτα. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ενημερωθούν και να συνηθίσουν οι καταναλωτές. Αυτό είναι το, πρώτο, το άλλο ερώτημα. Τρίτο, τελευταίο ερώτημα. Θέλουμε να προσθέσουμε την ετικετοθεσία στα ενδύματα. Οι πρόσθετες πληροφορίες που δίδονται μέσω διαδικτύου, όπως είναι στη ΣΥΠΑ το σύστημα, ένας ειδικό αριθμός, δεν άκουσα να τα αναφέρετε εσείς. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα για να δώσει βεβαιότητα στους καταναλωτές στη βιομηχανία. Μπορείτε να μας ενημερώσετε καλύτερα. Αν οι πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να δοθούν μέσω διαδικτύου για να μην δίνετε πληθώρα ε, πληροφοριών πάνω στο ένδυμα ή στον καταναλωτή που δεν ενδιαφέρεται. Ξέρω ότι σημειώνετε όλες τις ερωτήσεις. Θα ακούσουμε και άλλη ερώτηση η κυρία Γκέπχαρτ που εκπροσωπεί τον κύριο Σαλτεμόζα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαλτεμόζα έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα της ε, και μου ζήτησε να την ε, εκπροσωπήσω. Ε, πέρα από την ερώτηση που μόλις έθεσε ο κύριος Μάντες που αφορά την εναρμόνιση θα πρέπει να εξετάσουμε και ποιο θα είναι το κόστος της διαφορετικής επισήμανσης για 27 κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν γίνει υπολογισμός, να γίνει σωστός υπολογισμός και να μην υπολογίσουμε μόνο τη μία ε, πλευρά των δαπανών ε, χωρίς να υπολογίσουμε ε, την εξοικονόμηση που θα γίνει από κάποια άλλη πλευρά. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της εναρμόνισης από πλευρά τη προστασία των καταναλωτών και τη εσωτερική αγορά, θα πρέπει να είμαστε υπέρ εναρμόνισης στον τομέα αυτών, εάν θέλουμε να φροντίσουμε οι πολίτες να μπορούν να ψωνίζουν σε όλες τις χώρες της ε, εσωτερικής αγοράς. Αν ε, εγώ αγοράσω, για παράδειγμα, ένα προϊόν από το ίντερνετ, ε, θα, θέλω να γνωρίζω ότι θα μου κάνει το ρούχο και δεν θα χρειάζεται να το στείλω πίσω. Ε, αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Είπατε ότι το προαιρετικό σύστημα επισήμανσης για την φροντίδα δεν θα ήταν ε, ε, χρήσιμο για τους καταναλωτές. Μπορείτε να το στηρίξετε αυτό. Πρέπει να πω ότι μου έχει συμβεί στο μαγαζί μου έχει τύχει στο μαγαζί το, το, το προϊόν να γράφει ε, στεγνό καθάρισμα, ενώ η πολίτρια να μου λέει ότι δεν πειράζει και στο πλυντήριο μπορείτε να το βάλετε. Αυτό είναι σημαντικό θέμα, υποχρεωτικό σύστημα, ώστε να ε, περιγράφονται όλες οι δυνατότητες φροντίδας του προϊόντος. Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Ε, τρίτη ε, παρατήρησή μου. Δεν μου άρεσε πολύ η αιτιολόγησή σας γιατί θα πρέπει να εισάγουμε επισήμανση που έχει να κάνει με την χώρα προέλευσης. Ε, ήταν μάλλον προτεξιονιστική, προστατευτική η θέση σας. Ε, ερώτηση. Πόσο ψηλό είναι το ενδιαφέρον των καταναλωτών να έχουν για άλλους λόγους τις πληροφορίες αυτές. Για παράδειγμα, περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικοηθικά θέματα. Ξέρουμε, για παράδειγμα, <clears throat> ότι ε, κάποιοι ε, καταναλωτές δεν θέλουν να αγοράζουν προϊόντα από ε, χώρες όπου γίνεται χρήση εργατικού δυναμικού παιδιών. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κέπχαρτ. Εγώ θα έλεγα ότι στόχος μας είναι η εναρμόνιση και ταυτόχρονα όμως να πλουστεύσουμε την ετικετοθεσία. Επουδενή δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε τον καταναλωτή διότι και από τη μελέτη σας βλέπουμε ότι οι καταναλωτές θα ήθελαν να παραμείνει η ετικέτα ως έχει στην παρούσα μορφή. Θέτω αυτό το ερώτημα, διότι πολύ συχνά μου συμβαίνει η ετικετοθεσία είναι τόσο περίπλοκη, τόσο μακροσκελής, που δεν μπορεί να την καταλάβει ο καταναλωτής. Κατά άποψή μου πρέπει να δούμε και τις δύο πτυχές. Αν δεν παρατηρείται, δεν έχουμε ετικέτα γιατί θεωρείται άχρηστη ή δεν βάζουν την ετικέτα γιατί είναι δύσληπτη. Πολλές είναι πολύ λίγο ευανάγνωστες από τις ετικέτες έχουν κάποια ένδειξη, κάποια αναφορά περίπλοκη. Και χρειάζεσαι σχεδόν πτυχίο χημίας για να καταλάβεις μια ετικέτα, γιατί περιέχει τόσες λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο του υφάσματος. Η πολυγλωσία της ετικέτας. Θα ήθελα περισσότερες ευκρινήσεις πάνω σε αυτά που μας είπατε. Δεν νομίζω ότι οι καταναλωτέ ε, αρκούνται να έχουν μια τοκοθεσία τόσο μακροσκελή. Δεν του ικανοποιεί τόσο περίπλοκη ετικέτα και τόσο μακρό για να είναι όλε οι γλώσσε. Είναι ένα πλεονέκτημα για την επιχείρηση που δεν χρειάζεται να βάζει ξεχωριστέ ετικετέ κάθε, σε κάθε γλώσσα. Συμφωνώ με του προλαλήσαντε όσον αφορά το, τα μεγέθη, την ομοιομορφία των ε, μεγεθών. Είμαι Ιταλίδα και η χώρα μα είναι μία από τι πιο περίπλοκες χώρε για να μπορέσει κανεί να έχει ομοιομορφία όσον αφορά τα μεγέθη. Διότι για μα το ένδυμα είναι ένα είδο καλλιτέχνημα και είναι δύσκολο ε, να δώσουμε σαφή μεγέθη σε έναν Πικάσο, στα έργα του Πικάσο. Πιστεύω ότι ταυτόχρονα είναι θεμελιώδες να έχουμε μια ομομορφία για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διότι όποιο θέλει να πάει να αγοράσει κάτι, Dolce για καμπανά και αρμάνι, μπορεί να πάει επί τόπου και να τον βοηθήσει ο πολιτής. Όμως στην online πώληση δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τέλος, για τη χώρα προέλευσης, στην Ιταλία συζητείται αυτό περισσότερο από την Ευρώπη. Και στη χώρα μας, ακόμα περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη, είμαστε σε στάση αναμονής. Πιστεύω ότι και τα θεσία δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι, είναι, ότι η χώρα προέλευσης είναι η τελευταία χώρα στην οποία γίνεται τελευταία κατεργασία. Διότι αυτό είναι παραπλανητικό για τον καταναλωτή. Αν παράγω εγώ ένα ύφασμα παράγω ένα ύφασμα στην Κίνα, το μεταφέρω στην Ιταλία και βάζω το zip και τα κουμπιά και λέω είναι made in Italy, τότε αυτό δεν είναι η σωστή έννοια της χώρας προέλευσης. Το ερώτημά μου είναι, χρειάζεται να αναλύσουμε την ανεχνευσιμότητα του προϊόντος ή την ανεχνευσιμότητα. Ποια περάσματα πρέπει να αναφέρονται για να καταλήξουμε σε ένα made in που θεωρείται κατασκευασμένο το ε, αντικείμενο. Για τη χώρα προέλευσης, αυτά που μα είπατε, δεν νομίζω ότι είναι πολύ το ιδεώδε επιχείρημα. Διότι η χώρα προέλευσης καμιά φορά είναι, ε, δημιουργεί συνέστημα ασφάλεια. Η προέλευση προϊόντος δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, αλλά είναι και, δίνει και μια ασφάλεια, διότι σε κάποια προϊόντα που λέγονται Made in China στην Κίνα δεν χρειάζονται συγκεκριμένες δοκιμές που όμως απαιτούνται για τα προϊόντα παράγονται στην Ευρώπη. Οπότε είναι και θέμα ασφαλείας ε, και εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλερ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ έχω αρκετές ερωτήσεις. Καταρχήν ε, θα ήθελα να μάθω γιατί Περιγράψατε εσεί τα σημεία κίνηση, αλλά ένα από τα σημαντικότερα για μένα είναι ότι Πρόκειται για τεχνική πρόταση ώστε να καλύψουμε νέες ουσίες και ο κίνδυνος ε, με την οδηγία αυτή είναι ότι αν συμπεριλάβουμε υπερβολικά πολλά στοιχεία δεν θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Ιδιαίτερα η χώρα προέλευσης ε, θα δυσκολεύσει πολύ την όλη υπόθεση και ε, τα μειονεκτήματα μιας τέτοια οδηγία ε, που ε, πιθανόν να κολλήσει ε, στο Συμβούλιο δεν έχουν ληφθεί επαρκώ υπόψη. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνο καθυστέρηση. Όσον αφορά τα επιμέρους σημεία που αναφέρατε, αναφέρατε τις χημικές ουσίες. τα αλλεργιογόνα μου λείπουν εδώ. Θα Χαίρομαι που αναφέρεστε στην ανοτεχνολογία, την REACH κλπ. Αλλά αυτό που λείπει είναι οι αλλεργιογόνες ουσίε το, οποίο αφορά, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολλούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ηλεκτρονική επισήμανση, βρίσκω πολύ θετικό ότι αναφέρεστε στο θέμα της προστασίας δεδομένων, αλλά επίση ε, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η χρησιμότητα ε, πιο, πιο καθαριστήριο κοιτάει στο ίντερνετ πριν ε, ε, καθαρίσει ένα ρούχο. Ε, ουσιαστικά εδώ μετακυλούμε στον καταναλωτή την ευθύνη η οποία ανήκει στο, στην βιομηχανία. Δεν θα πρέπει στο ίντερνετ να υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχουν πάνω στο ένδυμα. τα υπόλοιπα ήταν αρκετά σαφή. Η, με ενδιαφέρει δηλαδή η εφαρμογή συστήματο για τι αλλεργιογόνε ουσία και η χρήση τη ηλεκτρονική επισήμανση. Και ακόμα. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα των οδηγιών φροντίδας. Ε, φυσικά είναι σημαντικό αυτό για τον καταναλωτή ε, όταν ε, δίνει στο καθαριστήριο ένα έντυπα διότι αν ε, το καθαριστήριο ε, δεν φροντίσει σωστά το ρούχο ε, ο καταναλωτής δικαιούται αποζημίωση. Δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και κάποιες απαντήσεις ίσως θα πρέπει να δοθούν αργότερα. Ήθελα να δώσω όμως τη δυνατότητα στα μέλη να θέσουν τις ερωτήσεις. Η κυρία Μακλάρκεν. Ευχαριστώ για την παρουσίαση τη μελέτη και των πολισμάτων τη μελέτη. Στα Ανατολικά Μίτλαν, στην περιοχή μου, είχαμε υπέροχη κλωστοϊφαντουργία Πολ Σμιθ στο Νόντιχαμ και δυστυχώ δεν είναι ποιόν τα πράγματα όπω ήταν. Παρόλο που υπάρχει ακόμα η κλωστοφαντουργία σε θύλακε. Αλλά όπω με πολλά ζητήματα που έχουμε συζητήσει, θέλουμε σωστή ισορροπία. Να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία και να προστατεύσουμε και του καταναλωτέ. Και καλό η ετικέτα να είναι σαφή. Να λέει τα πάντα όσα θέλει ο καταναλωτής κυρίως όσον αφορά τα λεριογόνα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, μην υπερφορτώνουμε την ετικέτα με πολλές πληροφορίες γιατί μπερδεύεται ο καταναλωτής. Και είναι βάρος και για τη βιομηχανία. Πρέπει να επικεντρωθούμε επί των ουσιαστικών στοιχείων. Και ποιες πληροφορίες πρέπει να διατίθεται τους καταναλωτές για να είναι πολύ ικανοποιημένοι από το προϊόν τους οι καταναλωτές. Αλλά μην βαρύνουμε υπερβολικά τη βιομηχανία και αυξάνουμε υπερβολικά το κόστος. Ερώτηση συνομιλήσατε με ενός καταναλωτών. Τους ρωτήσατε αν είναι πρόθυμοι οι καταναλωτές να πληρώνουν περισσότερα για να έχουν αυτές τις πληροφορίες. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κανονικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για ένα μέγεθος που ταιριάζει όλα. Και αυτό δεν λειτουργεί καθόλου όμως τελικά. Πολύ σύντομο ερώτημα. Κύριε Τιανταφυλλίδη, θέλετε να πάρετε το λόγο. με Πρόεδρε. Ο κ. Σαλβίνη θέλει να μιλήσει, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα. Ναι, για πέρα από αυτά που άκουσα, να πω ότι πρέπει να αποφύγουμε να γίνονται βιβλία πλέον αυτά και όχι ετικέτες. Πολύ εξειδικευμένε ετικέτες που ενδιαφέρουν κανέναν. Όμως όσον αφορά την Ιταλία, και όχι μόνο, είναι θεμελιώδους σημασία. Αφάνταστο να συζητάμε μια ετικέτα που να μην αναφέρει τη χώρα προέλευσης. Πρώτης ύλες, επεξεργασία, κατεργασία. Να ξέρουμε τα ποσοστά των χημικών συστατικών θα μπορούσε να είναι κάτι ε, ενδιαφέρον για τους ειδικού, αλλά όχι για την κυρία που αγοράζει κάτι στην υπεραγορά. Χώρα κατεργασίας παραγωγής είναι θεμελιώδου σημασίας να αναφέρεται. Δεν συμμερίζομαι τις παρεμβάσεις κάποιων συναδέλφων που λένε ότι κάνουμε τα πράγματα πολύ περίπλοκα ε, και να κάνουμε κάτι που και δεν συμφέρει να κάνουμε κάτι που βολεύει όλους αλλά δεν σε κανέναν. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα όσον αφορά την κατασκευή του προϊόντος. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ξέρω ότι καθυστερήσαμε και έχουμε και ακρόαση στις 10.30. Να δώσω στην κυρία Κινμόσεβιτς κάποια λεπτά. Δεν περιμένω να απαντήσετε στα πάντα. Ίσως γραπτός μπορείτε να μας στείλετε κάποιες απαντήσεις, αλλά ίσως κάποια βασικά ερωτήματα μπορείτε τώρα να τα απαντήσετε. Απάντηση ναι, με τα χαρά σας στείλω γραπτή, γραπτές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, το κόστος για την ετικέτα που αναφέρει πώς προσέχει κανείς το προϊόν. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα τέλη που καταβάλουν στις φορές τη Ginatex. Χρειάζεται αναδιπραγμάτευση με τη Ginatex ποια τέλη πρέπει να καταβάλλονται εάν θέλουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα. Όσον αφορά τις πωλήσει, την ιστοσελίδα μα του διαδικτύου για την εναρμόνιση, το εξετάσαμε και τι βρήκαμε. Ότι οι πληροφορίες που χορηγούνται μέσω του διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν συμπληρωματικές αλλά δεν μπορούν να διατεθούν αυτόνομες, διότι δεν έχουν όλοι οι καταναλωτές στη διάθεσή του το διαδίκτυο και δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιούν. Άρα στο σημείο πώληση χρειάζονται καμιά φορά οι πληροφορίες, αν είναι σε ένα κατάστημα δεν είναι πάντα εφικτό. Τώρα όσον αφορά τη χώρα προέλευσης, να ξεκαθαρίσω. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται η διοργάνωση εχνευσιμότητα του ενδύματο. Αναφέρομαι στην τρέχουσα πρακτική. Η χώρα προέλευση θεωρείται ότι είναι η τελευταία χώρα στην οποία το ένδυμα άλλαξε σημαντικά. Αυτό ίσως να μην αρκεί για τους καταναλωτές σαν πληροφορία, διότι όπως είπατε μερικοί από εσά σωστά θα θέλουν να ξέρουν αν το ένδυμα ή κάποια κομμάτια έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Οπότε υπάρχουν πιθανότητε αυτά που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα να μην συμμορφώνονται με την νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Για τα αλλεργιογόνα αναφέρουμε στη σελίδα 18 κάποια πράγματα. Αναφερθήκαμε και σε αυτό το θέμα. Τώρα, κατά πόσο οι κατανοητές θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για να έχουν στη θέση τους πληροφορίες. Αυτό ισχύει για τα χημικά, διότι αφορά την υγεία των καταναλωτών αλλά ίσως να μην αρκεί. Ίσως χρειάζεται να εξεταστεί διεξοδικότερα η ισχύουσα νομοθεσία. Και συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι οι καταναλωτές δεν θέλουν βιβλία, δεν θέλουν τεράστιες ετικέτες που δεν καταλαβαίνουν. Είναι υπερβολικό για αυτούς και δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνω τις πληροφορίες. Συμφωνώ ότι χρειάζεται προτεραιότητες στις πληροφορίες που χορηγούνται. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, που ήρθατε. Είναι πλούσια πηγή πληροφοριών η έκθεση. Αυτό ήταν και αρχικό σκοπός. Αν θα μπορούσατε να επανέλθετε επί κάποιων κρισίμων θεμάτων, θα μας βοηθούσε πολύ στη δουλειά μας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ή να κλείσουμε. Βλέποντα το χρόνο, θα ζητήσω από τους σκιώδους συζητητές για την επόμενη συνεδρίαση να δούμε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε και τις πρώτε πληροφορίε ταυτόχρονα και νομίζω ότι έληξε το θέμα διότι πρέπει να βιαστούμε. Πρόεδρος. Η κυρία Κιλμόσορβιτ, ίσω μπορεί να έρθει και στη συνεδρίασή σα και να γίνει πιο εκτενή συζήτηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε άλλη παρουσίαση, σε δύο άλλε μελέτε. Θα μα στριμώξει κάπω ο χρόνο. Θέλουμε να εστιαστούμε στην παρουσίαση. Η κυρία Ρούλε, που είναι διότι είναι δικές της μελέτες και οι δύο. Βγήκε. Εδώ είναι. Αν είναι έξω κυρία Ρούλε, ας τη φέρουμε. Έχουμε αναθέσει δύο μελέτες για τις δημόσιες προμήθειες. Η πρώτη αφορά τις συνέπειες της ε, συνθήκης της Αβώνας, τον αντίκτυπο της συνθήκης της Αβώνας ε, όσον αφορά ε, τις κρατικές προμήθειε. Η κυρία θα ασχοληθεί με αυτό. Και μετά έχουμε αυτό για την ανάθεση, για τι εκχωρήσεις. Η δόκτωρ Αν Κάρλιν Σάιντλερ θα αναφερθεί στο θέμα. Και οι δύο α, από το Φλίτζα Τεκαζέλε, την υπηρεσία αυτή, θα καλέσουμε καθέναν από εσάς θα δούμε διαδοχικά τις παρουσιάσεις και μετά θα υποβληθούν ερωτήσεις. Λόγω χρονικών περιορισμών, επειδή ακολουθεί ακρόαση, οι συγητέ ίσως να ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί σας αργότερα για περαιτέρω συζητήσεις. Ε, Δόκτωρ Ριζαν αν μπορεί να ξεκινήσει με τη δική της παρουσίαση, πρέπει να έχει τα αντίγραφα αυτών, συνάδελφοι, και είναι κακή εναρμόνιση αυτή να φαίνονται όλες οι εκθέσεις να έχουν την ίδια μορφή. Καλύτερο θα ήταν να έχουμε κάποιες γραφικές παραστάσεις, κάποιες εικόνες που να μας δίνουν κάποια εικόνα για το περιεχόμενο. Λοιπόν, είναι το εξώφυλλο παρόμοιο, αλλά το περιεχόμενο είναι διαφορετικό. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με μια σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων μας όσον αφορά τα ερωτήματά σας. Ετοιμάζοντας την παρουσίασή μας όσον αφορά τις επιπτώσεις της ηθίκης της Λισαβόνας στις δημόσιες συμβάσεις, αναλύσαμε πρώτα αλλαγές όσον αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Είναι κάπως διαφορετικό το θέμα το κατά πόσο υπάρχουν στη διαδικασία διαφορές εξαιτία της συνθήκης της Λισαβόνας. Αναλύουμε λοιπόν την κατάσταση κατά πόσο υπάρχει αρκετή ασφάλεια όσον αφορά τους ε, συμβαλόμενους. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, κυρίως όσον αφορά το άρθρο 3. Γιατί επικεντρώνεται η κοινότητα στο θέμα της ελεύθερης αγοράς, αλλά τονίζει και όλα τα μέτρα ανταγωνισμού. Νομίζω ότι εδώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι πειράζεται το θέμα των δημοσίων συμβάσεων και έχει υπάρξει και κριτική με την έννοια ότι ο ανταγωνισμός τελικά δεν προσαρμόζεται απόλυτα στο καθήκον που θα έπρεπε να έχει για τις διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις. Ο νέος ορισμός διευρύνει τους στόχους της Ένωσης και αντιστοιχεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη κάπως και κοινωνικές πτυχές. Όμως η νέα διατύπωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, ότι δηλαδή η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά μένει στο περιθώριο. Το άρθρο 119 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το, το πρωτόκολλο των 27 λέει ότι η προστασία των συστημάτων αγοράς για τον ελεύθερο ανταγωνισμό παραμένει ένα κεντρικό στοιχείο. Αυτό πρέπει να το δούμε και σε σχέση με όλα τα μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις. Κατά τη γνώμη μας, μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι η αναγνώριση των τοπικών και των περιφερειακών ε, αυτοχειριστικών μονάδων σε σχέση δηλαδή με τις υπηρεσίες κοινοφελών υπηρεσιών κυρίως. Τα περισσότερα πράγματα τα αναλαμβάνουν οι τοπικές δικήσεις των κρατών μιλών. Η συζήτηση συνεχίζεται για χρόνια πώς δηλαδή να λύσουμε την ελευθερία στις δημόσιες συμβάσεις και από την άλλη μεριά την ανάγκη των ε, τοπικών αρχών να αποφασίζουν από μόνες τους για το πώς θα φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Οι τοπικές αρχές συχνά διαμαρτύρονται για το ότι οι διαδικασίες των δημοσίων ε, ε, συμβάσεων τις εμποδίζουν να κανονίσουν τα πράγματά τους από μόνες τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Οι αλλαγές, πρέπει να σημειώσουμε, ότι Ε, έγιναν λαμβάνοντας υπόψη όσο γινόταν περισσότερο και τις ανάγκες των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές λοιπόν θέλουν να μπορούν να αποφασίζουν για ε, τα καθήκοντά τους όταν για παράδειγμα πρόκειται για συνεργασία δημοσίου-δημοσίου. Περισσότερες δυνατότητες λοιπόν για τις τοπικές αρχές προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται ήδη από την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η περίπτωση Κοντιτέλ, για παράδειγμα, όπου οι δημόσιες αρχές, ε, είπε το δικαστήριο, μπορούν να χρησιμοποιούν τους πόρους τους και μπορούν να το κάνουν και σε συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές. Η απόφαση αυτή Κοντιτέλ βασίστηκε σε συγκεκριμένη νομολογία όσον αφορά την in-house εξαίρεση. Και έχουμε και την άλλη περίπτωση, την Stadt Heringung Hamburg, με νέες εξαιρέσεις και με μια νέα έννοια που βασίζεται όχι σε τυπικές αρχές, αλλά σε μια νέα προσέγγιση που στηρίζεται πάλι στην, στο καθήκον της αρχής. Άλλο ένα στοιχείο που δείχνει πώς αλλάζουν τα πράγματα με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα γίνονται συζητήσεις για το ποιες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται για να μπορεί να υπάρχει εξαίρεση στον τομέα της συνεργασίας δημοσίου-δημοσίου. Οι προϋποθέσεις είναι ότι μόνο δημόσιες αρχές εμπλέκονται, ότι ο χαρακτήρας της ε, συμφωνίας πρέπει να είναι συνεργασία, πρέπει να υπάρχει αμοιβή και η συνεργασία βασίζεται στην επίτευξη στόχων υπέρ του κοινού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης εδώ να σημειώσουμε ότι δεν πρέπει οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να υποφελούνται ε, μία ιδιωτική επιχείρηση σε βάρος μιας άλλης. Από πλευράς διαδικασίας. Φυσικά η πιο σημαντική πτυχή είναι η αναγνώριση του περιφερειακού και του τοπικού ε, επίπεδου για την επικουρικότητα. Σε τομείς όμως που έχουν να κάνουν με αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή αυτή της επικουρικότητας περιορίζεται στον έλεγχο των ορίων αρμοδιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί όσον αφορά τις υπηρεσίες της κοινοφελής και εδώ είναι σε ένα βαθμό στο τοπικό επίπεδο και υπάρχει μια κάποια αλλαγή στη διατύπωση του άρθρου 14 ώστε να καλύπτει το θέμα της ρύθμισης. Βέβαια δεν είναι μια ευρεία αρμοδιότητα, οπότε δεν πρέπει να υπάρχουν ανησυχίες. Τωρινές διατάξεις. Οι νέες διατάξεις οδηγούν σε τροποποίηση της ερμηνείας της οδηγίας, της ήδη υπάρχουσας οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις νέες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έτσι υπάρχει μια νέα ερμηνεία όταν έχουμε να κάνουμε με μια σύμβαση επαμοιβή σε αντίθεση με μια συνεργασία που μπορεί να εξαιρείται. Έπειτα οι αλλαγές ανοίγουν το δρόμο σε δυνατότητες για τον νομοθέτη να επιλέγει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στον τομέα των κοινωνικών κριτηρίων μπορεί να οδηγηθούμε σε θέματα αξιολόγησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ε, ε, στόχοι που έρχονται σε αντίθεση ένας με τον άλλον. Είπαμε ότι υπάρχει ενίσχυση του ρόλου των τοπικών ε, δικήσεων. Επιτέχουμε τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Εδώ οι αλλαγές επιβεβαιώνουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Τώρα η χρήση των κοινωνικών κριτηρίων διευκολύνεται στο μέλλον. Όμως δεν είναι εντελώ ξεκάθαρο ποια θα είναι τα όρια. Συμπέρασμα. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι αυτός που ασχολείται με τις ε, δημόσιες συμβάσει. παραμένει σε αβεβαιότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια. Εδώ θα βοηθούσε πάρα πολύ να είχαμε μια ανακοίνωση για ερμηνεία, έτσι ώστε γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, όπως έχουμε και για τα περιβαλλοντικά κριτήρια, να ξέρουμε ποια είναι τα, τα περιθώρια κλπ. και στα κοινωνικά κριτήρια. Όσον αφορά τώρα την ε, διακοινωτική συνεργασία, και εδώ παραμένω βεβαιότητες για τις δυνατότητες και για τα όρια που μπαίνουν σε νέες δυνατότητες που ανοίγουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τι να κάνουμε με αυτές τις βεβαιότητες. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια ώστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προχωρήσει με αποφάσεις και έτσι να υπάρξει νομολογία για τα συγκεκριμένα όρια για ένα σωρό θέματα. Στο μεταξύ, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει δισταγμός από πλευράς της κοινότητας για λύσεις συνεργασίας ε, όσο οι αποφάσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε κατευθυντήρια γραμμή θα βοηθούσε, είτε πρόκειται για ανακοίνωση για ερμηνεία των αποφάσεων, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και αν υπάρξει τροποποίηση στη συνέχεια της οδηγίας που θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτούς που αποφασίζουν για δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τόσα μας είπατε. Θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Ακολουθεί όμως η ακρόασή μας και οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες για την ακρόαση άκουσαν την παρουσίασή σας και αυτό προσθέτει αξία. Διότι η πρώτη σύνοδος, το πρώτο τμήμα ε, της ακροάσης έχει τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που καλύπτει το κενό». Και το θέμα είναι κατά πόσο αυτός είναι ένας τρόπος σωστός για να αναπτύξουμε τον τομέα αυτών των ε, κρατικών, ε, κρατικών προμηθειών μπορείτε να επεκταθείτε αργότερα. Έχουμε δεύτερη μελέτη όσον αφορά τις εκχωρήσεις, αναθέσεις που διασυνδέεται με αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα καλέσω την κυρία Αν Κάρολιν Σάιτλερ να κάνει την παρουσίαση και λειτουργούν και τα συστήματα, οπότε θα φαίνονται και οι διαφάνειες στην οθόνη. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να μπορέσω να παρουσιάσω τα απορίσματα της μελέτης μας και θέλω να αναφερθώ στις εκχωρήσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έγιναν ε, πολλές συζητήσεις που ξεκίνησαν το 1971 ψηρά ετών κατά πόσο χρειάζεται νομοθετική δράση στο τομέα αυτών κυρίως όσο μιλά την αυξημένη χρήση των εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά καταρχάς στον ορισμό των εκχωρήσεων. Έχουμε ανάθεση έργων. Τι εννοούμε. Σύμβαση παρόμοιου τύπου όπως για δημόσια έργα με μια διαφορά. Ο... Είναι δικαίωμα εκμετάλλευση του έργου, αυτό που χορηγείται, ή δικαίωμα συλλογή πληρωμών, ίσπραξη πληρωμών. Έχω μια εικόνα, παράδειγμα κατασκευή και η λειτουργία σε δρομικής γραμμής. Η ίδια είναι η εκχώρηση. Μετά στην άλλη περίπτωση έχουμε υπηρεσίε που παρέχονται στη δεύτερη περίπτωση. Η λειτουργία ενός ε, τόπου αναψυχής, τοπικής αυτοδίκησης. Και το κοινό πληρώνει και έτσι αποπληρώνεται το έργο που τα χρήματα πληρώνει το κοινό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο ορισμός είναι πάρα πολύ ευρύς. Και ποια είναι η συνέπεια. Νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τις εκχωρήσεις αυτές. Συντάσσοντας το έγγραφο, τη μελέτη, διερωτηθήκαμε γιατί πρέπει να εντάσσονται αυτές οι αναθέσεις σε συγκεκριμένο καθεστώς. Δεν καταλήξαμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για αυτές τις ε, αναθέσεις. Για την πρώτη οδηγία περί υπηρεσιών έγινε κάποια πρόταση. Προτάθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις για τις αναθέσεις και αναθέσεις έργων πιο συγκεκριμένα. Διαγράφησαν όμως από το Συμβούλιο. Γιατί? Υπήρχε μεγάλη διαφορά εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις εκχωρήσεις σε αυτό τον τομέα. Αυτό ήταν ο μόνος λόγος που βρήκαμε για τη διαγραφή. Ποια είναι η υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε τον ορισμό της οδηγίας 2004-18 ΕΟΚ για του δημόσιου τομέα. Έχουμε και τον κανονισμό για τις ε, δημόσιες μεταφορές που υπάρχουν κανόνες για την Έχουμε τις αρχές τη συνθήκης εν γέννη και έχουμε την ερμηνευτική ανακοίνωση. Υπάρχουν πολλοί κανόνες. Είναι εμβαλωματικέ λύσεις, ένα μοσαϊκό κανόνων. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Ποια είναι η συνέπεια. Υπάρχει πρόβλημα διάκρισης δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεων, εκχωρήσεων. Δεν υπάρχει σαφής διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Κάθε κράτος μέλος ακολουθεί ειδικού του κανόνες. Δεν υπάρχει ομοιομορφία όσον αφορά την εφαρμογή των εκχωρήσεων. Πήγαμε στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και είπαμε μήπως βρούμε κάποια κατεύθυνση από την ομολογία. Όσον αφορά τις εκχωρήσεις αναθέσεις έργων, δεν βρήκαμε κάποια υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε και μπήσε λεπτομέρειε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπήρχε κάποια αναφορά σε κάποιε υποθέσει. Στο μέλλον ίσως τοποθετηθεί το δικαστήριο σε μελλοντικέ υποθέσεις, εξεπώνηθηκαν κάποιες γνωμοδοτήσεις αλλά δεν υπάρχει νομολογία του δικαστηρίου ακόμα για τις αναθέσεις έργων. Διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τις αναθέσεις υπηρεσιών. Υπάρχουν πάρα πολλέ υποθέσεις, κυρίως διάκριση μεταξύ δημόσιων συμβάσεων και ε, αναθέσεων. Όταν είδαμε τις υποθέσεις, τι ανακαλύψαμε. Δεν υπάρχει σαφής διαφορά, κυρίως όσον αφορά το δικαίωμα εκμετάλλευσης υπηρεσίας, αν θυμώ τον ορισμό. Και το δικαστήριο προσέθεσε λεπτομέρειες στην περίπτωση Πάκιν Μπρίξεν, είπε το δικαίωμα εκμετάλλευση υπηρεσία πρέπει να περιέχει ανάληψη κινδύνου για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Άρα εννοείται ότι ε, ε, λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος για την χορήγηση υπηρεσία. υπηρεσίας. Είχαμε πρόσφατη υπόθεση, ο Ιντουρκ Τεχνίρ και ο οι Υπήρχαν διαφορετικέ προσεγγίσεις που ακολουθηθήκαν στις δύο υποθέσεις όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου. Δηλαδή ο εμπορευόμενος πόσο κίνδυνο πρέπει να αναλάβει. Ίσως διότι διαφορετικοί φορείς του δικαστηρίου ασχολήθηκαν, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σαφής κανόνας Πώς χορηγείται η ανάθεση, ποια διαδικασία. Το δικαστήριο είπε εφαρμόζεται μόνο, εφαρμόζονται μόνο οι γενικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό όμως, τι σημαίνει εφαρμογή των γενικών αρχών. Βλέποντας όλες τις πηγές και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τους νομικούς κανόνες κλπ, Δημιουργείται ερωτηματικό. Χρειάζεται κάποια δράση στον τομέα αυτό των αναθέσεων. Θα μπορούσατε να δηλωτηθείτε αν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Ίσως η νομική αυτή η αβεβαιότητα οδηγήσει σε μείωση ανταγωνιστικότητας, απώλεια ανταγωνιστικότητας και έλλειψη ασφαλείας όσον αφορά τις επενδύσεις. Υπάρχουν πολλές επιλογές του τι θα μπορούσε να ρυθμιστεί στον τομέα αυτό πού θα έπρεπε να αναλυφθεί η δράση. Μια επιλογή θα ήταν ερμηνευτική ανακοίνωση. Ίσως μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αυτό δεν αρκεί, αυτή η ερμηνευτική ανακοίνωση, διότι συνοψίζει και επεξηγεί υφιστάμενους νόμους και νομολογία. Και ίσως όμως δεν υπάρχει βιώσιμη ασφάλεια δικαίου τρόπος. Άλλη επιλογή. Ειδική νομοθεσία για όλα τα έργα που αφορούν μετάθεση κινδύνου. Αυτό θα επέλυε το πρόβλημα που ίσως στην αρχή της διαδικασίας είναι δύσκολο να γνωρίσει κανείς στην αρχή της εκχωρήσεως ποιο είναι το πιθανό αποτέλεσμα. Λεπτομερέστερο καθεστώς ίσως να μην χρειάζεται διότι έχουμε ήδη διαδικασίες που προβλέπουν οι οδηγίες και ίσως να, οι προβλέψεις της οδηγίας να αρκούν για τις αναθέσεις άλλη λύση, ξεχωριστή νομοθεσία για αναθέσεις που είναι εκτός του πλαισίου της οδηγίας. Ποιο θα ήταν το πρόβλημα. Θα υπάρχει πρόβλημα ορισμού που ίσχυε σε άλλες περιπτώσεις και ήταν το βασικό πρόβλημα. Διάκριση μεταξύ δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεων. Άλλο ερώτημα. Χρειάζεται νέα διαδικασία. Χρειάζονται και άλλες ρυθμίσεις και άλλοι κανονισμοί για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη βεβαιότητα. Αυτά είναι όλα ερωτήματα που θα πρέπει να τεθούν. Άλλη δυνατότητα, τρίτη δυνατότητα. Να ρυθμίζονται αυτές οι αναθέσεις στα πλαίσια της ισχύουσης οδηγίας και να χρησιμοποιούνται όμως να εξασφαλιστεί ότι οι φυστάμενες διαδικασίες ταιριάζουν αυτόν τον σκοπό. Είναι οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι οι δύο διαδικασίες. Ποιο θα ήταν το όφελος. Δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα διάκρισης. Σαφείς κανόνες, ένα κείμενο. Εν τη αυτή περίπτωση. Ένα επιχείρημα κατά. Θα άλλαζαν οι ισχύουσες πρακτικές. Έτσι και θα υπήρχε ασυνέπεια όσον αφορά την εφαρμογή και εχθρό τη εκ μέρους των αγοραστών ενδεχομένως. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια επιχειρήματα να αποφασίσετε τι πρόβλημα πρέπει να ρυθμιστεί, να μην ρυθμιστεί, αν χρειάζεται σε μελλοντικές υποθέσεις να υπάρξει ρύθμιση ή όχι. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Και οι δύο παρουσιάσεις υπήρξαν σαφέστατες και υπογράμμισαν τα βασικά ζητήματα. Η κυρία Ρούλε ξέρω ότι ασχολείται με αυτά τα θέματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε την ακρόασή μας εγκαίρως. Έχουμε ένα τέταρτο περίπου για κάποια σχόλια από τα μέλη. Ίσως θα σας ζητήσουμε να πανέλθετε για κάποια από τα θέματα. Ίσως η κυρία Ρούλε μπορεί να αναφερθεί στο θέμα. Καλωσορίζω και τον κύριο Βλάσεκ που είναι εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής ευπρόσδεκτος. Πολλά από τα θέματα της συνθήκης αφορούν, ε, μάλλον συνεπάγονται, ε, η νέα συνθήκη συνεπάγεται μεγαλύτερη επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυρία Ρούλε να σχολιάσει, ο κύριος Βλάσεκ ίσως θέλει να σχολιάσει τώρα, παρόλο θα μιλήσει και αργότερα και θα ακούσουμε και άλλους σκιώδεις που είναι παρισταμένοι. Ο κύριος Έγγελ είναι εδώ. Πού είναι ο κύριος Έγγελ? Να, στη δεύτερη σειρά είναι. Α, δεν τον είδα. ο κύριος Έγκλ, κύριε Βανιού, ο Κρόιτσμαν, εγώ είμαι εδώ, είμαι σκιώδης για την ομάδα μου και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ, οπότε ξεκινάμε. Είχα τη δυνατότητα να διαβάσω την ε, μελέτη σας, αν και την έλαβα σχετικά αργά. Πρόλαβα όμως να τη διαβάσω και ε, πρόκειψαν κάποιες ερωτήσεις. Ε, καταρχήν, όσον αφορά τις αποφάσεις που αναφέρετε, αναφέρετε αρκετές αποφάσεις του ΔΕΚ στην ε, μελέτη για τις ε, συμβάσεις παραχώρησης που βασίζονται στην ε, παλιά οδηγία του 1998. Μόνο δύο περιπτώσεις αναφέρονται στην νέα οδηγία του 2004. Όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, η νέα οδηγία είναι πολύ πιο σαφής από την παλιά και αυτό το ε, και το αναφέρει αυτό το ΔΕΚ ε, στο ε, σημείο 39 και 54 της απόφασης Eurovaser. Αναφέρεται στην μεταφορά του κινδύνου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει νομική αβεβαιότητα. Επίσης, ως προτιμητέα λύση ε, ε, είναι οι συμβάσεις παραχώρησης να συμπεριληφθούν ε, στην οδηγία για την ανάθεση έργων. Αλλά υπήρχε αντίθεση σε αυτό από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Γιατί δεν αναφέρετε τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου το 2004 κατά της λύσης αυτής. Θα ήταν χρήσιμο. Και Απόρρισα επίσης ε, γιατί λαμβάνεται σε ε, χαμηλό βαθμό υπόψη την ε, γαλλική συζήτηση που έχει γίνει για το θέμα. Αναφέρεστε στην γερμανική φιλολογία για το θέμα, στην αγγλική, αλλά... Μου φαίνεται ότι αυτή ακριβώς είναι η αποφασιστική σημασία συζήτηση για το θέμα αυτό. Γιατί το Κοινοβούλιο τότε δεν ήταν υπέρ της συμπερίληψης των συμβάσεων παραχώρησης ε, στην ε, οδηγία για την ανάθεση έργου, για να ε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας. Γι' αυτό αναρωτιέμαι σχετικά με τα, αποτελέσμα... με τα συμπεράσματά σας, αλλά μήπως μπορείτε να μας σχολιάσετε περαιτέρω. Όσον αφορά το πρώτο θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας και των συνεπειών στην, ε, στις δημόσιες προμήθειες. Έχω δύο ερωτήσεις λέτε ότι με τη Λισαβόνα έχουμε μια νέα κατάσταση η οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστεί νομικά. Απ' την άλλη, στο κείμενό σας, στη σελίδα 8, αναφέρετε την υπόθεση Κόντιτελ Μπραπάντ και αναφέρετε τις, ε, τα συμπεράσματα που ήδη έχει εξάγει ε, το ΔΕΚ από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει πράγματι νομικό κενό, δεν είναι σαφής νομική βάση. Έχουμε την ε, απόφαση Στάτβερ και Χάμπουργκ. Ε, προτείνεται στην, ε, στα εγγραφά σας μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Τι εννοείτε με αυτό η διαδημοτική συνεργασία, η συνεργασία ε, διαφόρων δημόσιων φορέων μεταξύ τους ε, θα ε, συμπεριλαμβάνονται στο μέλλον στην, στην, στις δημόσιες προμήθειες και αν ναι, γιατί δεν το λέτε και παρακαλώ να μου το εξηγήσετε αυτό περαιτέρω. Ευχαριστώ. Μπορεί να μην προλάβουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σήμερα. Κύριε Βλάσεκ, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με αυτά που, ήδη ακούσατε. Ο κύριος Έγγελ τότε. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά θέλω να επιβεβαιώσω, να τονίσω κάποια από τα πράγματα που είπε και η κυρία Ρούλε όσον αφορά αυτή την εκχώρηση έργου. Όσο δεν έχουμε το γαλλικό στοιχείο μέσα στην εικόνα, δεν έχει νόημα να μιλάμε για αυτές. Διότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία λογική ευρωπαϊκών εκχωρήσεων αν δεν λάβουμε υπόψη μας και την γαλλική λογική μέσα στην ευρωπαϊκή λογική ή αν δεν κάνουμε την ευρωπαϊκή λογική γαλλική λογική. Άρα είναι μια θεωρητική και ακαδημαϊκή φύσεως συζήτηση αυτή που έχουμε, όσο δεν διαθέτουμε και τα κύρια στοιχεία, που είναι η γαλλική πραγματικότητα, που ισχύει εδώ και 200 χρόνια περίπου. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βαρνιό, συμφωνείτε? Θέλατε το λόγο, δεν θέλατε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι, συμφωνώ. Οι δύο παρουσιάσεις που ακούσαμε και σας ευχαριστώ πολύ για αυτές, αντί να μου λύσουν ε, κάποιες απορίες, μου δημιούργησαν παραπάνω. Είναι αλήθεια, είπατε κι εσείς ε, σίγουρα αλλάζουν τα δεδομένα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζω ότι από νομικής άποψης θα έχουμε μια βάση, αλλά θέλω και ένα κείμενο που να στέκει. Και ο προλαλής σας ακριβώς γι' αυτό μίλησε. Στη Γαλλία βλέπετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτά και έχουμε αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες για να θέσουμε σε εφαρμογή τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο όλα αυτά. Πάλι καλά πάνε τα πράγματα, δεν έχω παράπονο. Πάντα υπάρχουν κάποια προβλήματα ορισμού, πάντα υπάρχουν κάποια προβλήματα αβεβαιότητας για τις επενδύσεις, γιατί βλέπετε δεν προβλέπονται τα πάντα από το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο Άρα χρειάζεται διευκρίνηση όταν πρόκειται για εθνικές περιφερειακές αρμοδιότητες και τι είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα τώρα μετά τη Λισαβόνα. Τα κριτήρια τώρα, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, νομικό κενό. Και είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον έτσι όπως εγώ βλέπω τα πράγματα, εγώ που βγαίνω σε Δήμο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κριτήρια. Γι' αυτό μιλάω για νομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί. Αυτά που ακούσαμε δεν νομίζω ότι καλύπτουν αυτό το κενό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα θέμα με ενδιαφέρει από αυτά που ακούσαμε στην παρουσίασή σας. Σε τι βαθμό η απόφαση του ΔΕΚ για το Αμβούργο έχει συνέπειες στην ελεύθερη αγορά. Από τη μία είπατε ότι η βασική αρχή είναι ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά στις δημόσιες προμήθειες. Από την άλλη, η Δήμοι προσπαθούν με νέες δομές να αποφύγουν τις, ε, τις ελεύθερες δημόσιες προμήθειες. Αυτή τη δομή βλέπουμε στην Γερμανία. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε τι βαθμό αυτή η αντίφαση, αυτή η αντίθεση η εσωτερική αγορά από τη μία και από την άλλη η απόφαση του ΔΕΚ όπου δίδεται η εντύπωση ε, ότι ε, υπάρχουν εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Πώς βλέπετε εσείς την αντίθεση αυτή. Νομίζω ότι μπορώ και εγώ να κάνω μια σύντομη παρατήρηση ως και ε, για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο στα αριστερά μου. Ιδιαίτερα με ενδιαφέραν οι παρατηρήσεις που κάνατε για κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που συζητήσαμε στα πλαίσια της οδηγίας του 2004 που στόχο είχαν να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτές τις πολύπλοκες συμβάσεις όπως είναι οι συμβάσεις παραχώρησης. Πρόκειται για δύσκολες συμβάσεις ε, κατά τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με άλλες αναθέσεις έργου και φαίνεται να υπάρχουν κάποια ευρύτερα θέματα ε, που προκύπτουν σχετικά με το πώς λειτουργεί ο ανταγωνιστικός διάλογος και κατά πόσο λειτουργεί με συνέπεια η νομοθεσία, διότι ένα από τα προβλήματα ήταν να τεθούν όρια η διαπραγμάτευση των, ε, αναθετουσών αρχών ε, με μια σειρά ε, υποψηφίων μέχρι κάποιο σημείο. Κάτι τέτοιο δίνει μεγάλη ευελιξία. Ε, κάποιοι θα λέγανε υπερβολική ευελιξία σε κάποιους τομείς, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να εξεταστεί αυτό που προτείνατε το αν η ευελιξία αρκεί για να καλύψουμε τις συμβάσεις παραχώρησης ε, και αν αυτό συνάδει με αυτά που είπαν νωρίτερα οι συναδελφοί μου. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ε, ποια βήματα, τι πρέπει να κάνουμε για να ελοποιηθούν έτσι που να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση στο βαθμό και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αναθέτουσες αρχές και επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις ρυθμίσεις και σε κράτη-μέλη που δεν επιβάλλουν την εφαρμογή των διατάξεων σε εθνικό επίπεδο. Και δεύτερο, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην αγορά και ποια μέτρα να ληφθούν για να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Uh, right. Well, um... Uh, Καλώς. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο για να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Θα κάνουμε όπως και με το προηγούμενο θέμα. Δηλαδή απαντήστε σε κάποιες και στις υπόλοιπες γραπτά. Δόκτωρ Σάλλον, Πρώτα, μήπως σύντομα παρακαλώ. Ε. Και μπορείτε να μείνετε και μετά, αν θέλετε, στην ακρόασή μας βέβαια. Θα απαντήσω στα γερμανικά. Μου φαίνεται πιο απλό. Καταρχήν, όσον αφορά την ερώτηση, σε ποια βάση έχει εκδοθεί η νομολογία του ΔΕΚ. Πράγματι, οι περισσότερες αποφάσεις έχουν εκδοθεί με βάση όχι τη νέα οδηγία, αλλά τον ορισμό των συμβάσεων παραχώρησης που υπήρχε πριν από αυτήν. Η νομική αβεβαιότητα προκύπτει ακριβώς από το σημείο τι είναι η μεταφορά κινδύνου, πόσο υψηλή θα πρέπει να είναι και στο θέμα αυτό δεν υπάρχει διαφορά στον, ανάμεσα στον νέο ορισμό και τον ορισμό που έχει χρησιμοποιηθεί νωρίτερα κατά την ε, έκδοση της νομολογίας του ΔΕΚ. Η όλη προβληματική δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα από εθνικά δικαστήρια για το πώς θα πρέπει να ερμηνευτεί ο ορισμός αυτός. Δεν έχει εισαχθεί περισσότερη βεβαιότητα με τη νέα οδηγία. Όσον αφορά το θέμα της πολιτικής συζήτησης Θέλουμε να αναλύσουμε την ε, νομολογία του ΔΕΚ και για να καταλήξουμε σε ε, νομικές διατάξεις, σε νομικές οδηγίες και νομίζω ότι ακριβώς αυτό κάναμε. Ε, όσον αφορά τον την τελευταία ερώτηση, τον ανταγωνιστικό διάλογο, την διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα προβλήματα που συναντάει η Γερμανία και άλλες χώρες μάλλον οι εμπειρίε που έχουν ε, τα κράτη-μέλη δεν είναι ε, πάρα πολλέ ε, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον έχει περισσότερη εμπειρία με τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να συνδυαστούν οι εμπειρίε. Σύντομα όσον αφορά τις ερωτήσεις για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρώτη ερώτηση, εάν στην ε, διαδημοτική συνεργασία υπάρχει ε, ανάγκη ε, για περισσότερη νομική βεβαιότητα όσον αφορά τις αποφάσεις του ΔΕΚ για την Κοντιτέλ Μπράπαντ και την Eurovaser. Με την ανάλυση των δύο αυτών ε, περιπτώσεων ε, προκύπτουν ε, κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε αναφέρει. Για παράδειγμα, η διάκριση ανάλογα με τον χαρακτήρα της συνεργασίας και το είδος της σύμβασης θα πρέπει να πούμε ότι το ΔΕΚ στην περίπτωση Στάτρα Χάμπουργκ έχει ξεφύγει κάπως από τον πολύ στενό ορισμό. Αυτό είναι χρήσιμο για όσους ε, ασχολούνται με τις ε, συμβάσεις αυτές. Όσον αφορά την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και την ε, και το να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Κατά τη γνώμη μας ε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας εδώ, αλλά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι πιο σαφή, πιο συγκεκριμένα, ώστε στον τομέα αυτών να μπορέσουμε να συνδυάσουμε καλύτερα τους στόχους της ε, Ένωσης. Όσον αφορά τη δυνατότητα διαδημοτικής συνεργασίας ε, και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ε, μια ε, σύμβαση όπου παρέχονται υπηρεσίες ε, με οικονομικό αντάλλαγμα ε, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας των δημοσίων προμηθειών άσχετα από το αν μιλάμε για δημόσιους φορείς. Δεν υπάρχει παρανόηση της νέας νομολογίας του ΔΕΚ Ήδη το ΔΕΚ έχει ε, καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται απλά για γενικό πράσινο φως ε, ε, οι δημοτικές συνεργασίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο συνεργασίας όπου υπάρχει μοίρασμα και των οργανωτικών μέτρων. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν εφαρμόζεται το δίκαιο που αφορά τις δημόσιες προμήθειες τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει η διάκριση και θα βοηθούσε την όλη πρακτική εάν είχαμε περισσότερη σαφήνεια στον τομέα αυτόν. Αν μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα, ε, κίνητρα για την συμμόρφωση με τους κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις θα είναι η τελευταία ερώτηση. Αυτός αποτελεί έναν από τους στόχους της νέας οδηγίας. Τίθεται όμως πάντα το ερώτημα τι κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Κατά τη γνώμη μας, από τις νέες διατάξεις δεν προκύπτουν σημαντικές τροποποιήσεις τώρα με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, η οδηγία για τα ένδικα μέσα αποτελεί κατά τη γνώμη μας σημαντικό βοήθημα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τις δύο θερμά για τη δουλειά σας πάνω στο θέμα αυτό και ε, θα, θα ήθελα να παραμείνουμε σε επαφή διότι η κυρία Ρούιλε και άλλοι έχουν ε, ερωτήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η κυρία Ρούιλε θα ζητήσει να συμμετάσχετε στη συζήτηση και ε, για τους προσκεκλημένους μας ε, που ήρθαν για την ε, ακρόαση. Τα έγγραφα υπάρχουν εδώ πέρα σε χαρτί, αλλά θα είναι διαθέσιμα και σε, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Και θα παρακαλούσα τις κυρίες να παραμείνουν και να ακούσουν τη συζήτησή μας. Να περάσω λοιπόν χωρίς διακοπή στην ακρόασή μας ε, που έχει να κάνει με τις ε, δημόσιες συμβάσεις ε, και τις νέες προκλήσεις που συνδέονται με αυτές. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες μας. Επειδή ξεκινήσαμε τη δουλειά μας στις 9 η ώρα, δεν είχα τη δυνατότητα να χαιρετήσω προσωπικά ε, το, το, τους εμπειρογνώμονες μας. Ε, ε, πρέπει να πω όμως ότι ε, δεν είναι ετούτη αίθουσα αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως για ακροάσεις, επειδή όμως είχαμε κάποια, κάποια θέματα διοργάνωση αυτή τη βδομάδα, αλλάξαμε αίθουσα, βρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα. Δυσκολεύομαι να δω και τα ονόματά σα ε, σε αυτή τη σφαιρική, σε αυτή την κυκλική αίθουσα. Είναι δύσκολο να βλέπω όλου. Παρακαλώ λοιπόν να δείξετε κατανόηση. Επίση, οι συνάδελφοι κάθονται σε κάπω ε, διαφορετικέ θέσει από ό,τι συνήθω. Να καλωσορίσω λοιπόν πρώτα του ε, εμπειρογνώμονε, του οποίου θα σα παρουσιάσω αργότερα. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω και πάλι και να ευχαριστήσω την Χάιντι Ρούιλε που βρίσκεται εδώ στα αριστερά μου είναι η συγγήτρια για το θέμα αυτό και τον κύριο Βλάσεκ, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, και τον κύριο Χάνσλικ που είναι ε, συντάκτης της νομοδότησης ε, ε, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, από τον οποίο θα ακούσουμε λίγα λόγια σε λίγο. Και έχουμε τον κύριο Βίνα από την Επιτροπή, από την Κομισιόν και εσάς σας έψαχνα, διότι δεν κάθεστε εκεί συνήθως. Ξέρω ότι έχουμε κάποιους εκπροσώπους από την Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά που παρακολουθούν στενά τις εργασίες αυτές και οι συμβάσεις παραχώρησης ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν στον κύριο Μπαρνιέ ε, σε μια ακρόαση πριν λίγο καιρό. Ο κύριο Μπαρνιέ εξακολουθεί να είναι μέλο τη επιτροπή μα ε, μέχρι να οριστεί επίσημα Επίτροπος. Ε, ο χρόνος μας πιέζει, θα χρησιμοποιήσουμε το ρολόι για τους ομιλητές ε, και ε, επειδή έχουμε μέσα σύγχρονε τεχνολογίε, θα βλέπετε το χρόνο μπροστά σας. Ε, δεν θα δυσκολευτείτε λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο. Θα παρακαλούσα την Χάιντι Ρούιλε να παρουσιάσει την ακρόαση. Υποσχέθηκε να μιλήσει για τρία λεπτά, οπότε θα δοκιμάσουμε το σύστημα μέτρησης του χρόνου με αυτήν. Κύριε Βλάσια, και εσείς τρία λεπτά θα έχετε. Θα παρακαλούσα λοιπόν να συμπιέσετε όσο γίνεται την παρουσίασή σας και κατόπιν θα ακούσουμε τις επιρρογνώμονες. Κίτρινοι φάκελοι υπάρχουν με αντίγραφα των διαφανειών. Ε, αυτά νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κυρία Ρούλη σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη για να δώσω και περισσότερο χρόνο στον κύριο Βλάσεκ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους ε, και τον πρόεδρο της Επιτροπής μας ε, που ε, κατέστησε δυνατή την σημερινή ακρόαση. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας ασχολείται εδώ και χρόνια με το θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Να σας θυμίσω ότι είχαμε την έκθεση Μακάρθη που ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής μας για θέματα εφαρμογής και επιβολής του νόμου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Είναι σημαντική έκθεση. Έχουμε την έκθεση του ε, Προέδρου μας, ε, κ. Χάρβορ, για την καινοτομία που έχει ε, Όλα αυτά ε, ε, μας οδηγούν στο ερώτημα γιατί ασχολούμαστε πάλι με το θέμα αυτό. Στην οικονομική ε, κρίση, σε οικονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντικό ο τομέα των δημοσίων προμηθών. 16 με 17% της οικονομίας καλύπτονται έτσι και οι εμπλεκόμενοι παραπονιούνται για το, για το μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να συμμετέχουν στις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις υπάρχουν ε, σημαντικές δαπάνες λόγω, νομικής, λόγω ανάγκης για νομικές συμβουλές αλλά και γενικά είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούσαμε ήδη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει επιπτώσεις στο θέμα της δημοτικής αυτοδιοίκησης και τον ρόλο των Δήμων. Αυτό που μας απασχόλησε ε, στο προ... Αυτό μας απασχόλησε καταρχήν και σύμφωνα με αυτό έχουμε ε, δομήσει την ακρόασή μας. Αναφέρθηκαν κάποιες ερωτήσεις όπως η Stadt Reinigung Hamburg και η Kotitel Brabant, η Eurovasser οι αποφάσεις αυτές του ΔΕΚ ε, μας οδηγούν στο ερώτημα εάν το ΔΕΚ ήδη έχει κλείσει τα νομικά κενά ή αν υπάρχει ακόμα ανάγκη ε, να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Ε, σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τις διαδημοτικές συνεργασίες, δηλαδή οι συνεργασίες μεταξύ δημοσίων φορέων, καθώς και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Public-Private Partnerships, PPP. Οι οδηγίες αυτές ε, δίνουν ε, την δυνατότητα ε, στις επιχειρήσεις να ψάξουν την οικονομικά πιο συμφέρουσα λύση, ε, να ληφθούν υπόψη και κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω και τη το ήπιο δίκαιο, το προαιρετικό δίκαιο που έχει σαχθεί τα τελευταία χρόνια το soft law το λεγόμενο, ε, που συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Την κυρία Ρούλε. Βλάσακ. Έχουμε και τις διαφάνειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο περίπλοκα πράγματα με τα οποία έχουμε να κάνουμε στην Ευρώπη επί του παρόντος. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι 16% του ετησίου ΑΕΠ όλων των χωρών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτέ, διότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα που να απειλούν την οικονομική μα ανάπτυξη. Οι δημόσιε συμβάσει λοιπόν δημιουργούν προβλήματα ε, σχετικά με την χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο, η συνοχή είναι ο τομέα όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί λένε ότι 11% του συνολικού ποσού που επιστρέφεται δεν πληρώνεται τελικά και ότι 80% των περιπτώσεων έχουν σαν κύριο λόγο ε, προβλήματα με την τήρηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πιο πρόσφατη εμπειρία μας δείχνει ότι οι δικαιούχοι δυσκολεύονται να εφαρμόσουν καλά τους κανόνες με τις δημόσιες συμβάσεις. Τα πιο συνηθισμένα λάθη όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων είναι η τήρηση των κανόνων όσον αφορά την προσφορά και οι διαχειριστικές αρχές τι λένε. Λένε τι κάνουν τελικά. Μειώνουν τις, ε, τα χρήματα που έχουν υποσχεθεί. Το πρόβλημα μπορεί να μην είναι τόσο πολύ το ότι δεν έχουμε νομικό πλαίσιο όπως θα έπρεπε, αλλά συχνά έχει να κάνει με την μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο ή την εφαρμογή των κανόνων από το επίπεδο το οποίο εφαρμόζει και τους κανόνες. Τι φταίει σε αυτό, ίσως δεν υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση, δεν υπάρχουν σωστές κατευθυντήριες γραμμές, ναι. Αλλά το βέβαιο είναι ότι πρέπει να είναι καλά γνωστή η νομοθεσία και τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την κατάρτιση ειδικών που να μπορούν να εφαρμόζουν τους κανόνες στις δημόσιες συμβάσεις. Πέρα από τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση κοινοτικών πόρων, οι Δήμοι πολύ συχνά διαμαρτύρονται και για την έλλειψη διαφάνειας. Υπάρχει αβεβαιότητα, γραφειοκρατία. Χρειάζεται διάκριση ανάμεσα στα δημόσια, στις δημόσιες συμβάσεις και ε, τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις, περιορισμοί που μπαίνουν στους Δήμους δυσκολεύουν τους Δήμους ή προβλήματα επίσης με τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Σε αυτούς τους τομείς οι δημόσιες αρχές δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν σωστά τους κανόνες. Θα έπρεπε λοιπόν να καθίσουμε και να κοιτάξουμε ποια είναι η άποψη των ειδικών και των οργανώσεων εκείνων που ασχολούνται με το νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό και είναι πολύτιμες ακροάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βλάσακ. Όντως, ευχαρίστω σαν ειδικό να σας έχουμε εδώ, ξέροντας ότι δουλεύετε πολύ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οπότε η άποψή σας είναι πολύτιμη για μας. Καλώς. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στους εμπειρογνώμονες που έχουμε καλέσει για την καλύτερη νομοθεσία και κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φτάνει για να καλύψει το κενό ερωτηματικό. Θα σας παρουσιάσω τους ειδικού. και ελπίζω να είσαστε όλοι εδώ και να πω σωστά τα ονόματά σας. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τον Ρομπ Χάν, ο οποίος εκπροσωπεί το Συμβούλιο Περιφερειών και Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε πολλή γνώση για το θέμα. Ο κύριος Βλάσακ πριν από λίγο αναφέρθηκε στην κατάρτιση και την εκπαίδευση των τοπικών αρχών για τις δημόσιες συμβάσεις. Μετά έχουμε τον Στέφανο Ροντρίγκε, τον καθηγητή. Α, είσαστε με τη σειρά. Ωραία. Που είναι δόκτωρα στο κοινοτικό δίκαιο. Οικονομικό δίκαιο επίση στο Παρίσι, που έχει δημοσιεύσει πολλά πράγματα στον τομέα των ε, δημοσίων υπηρεσιών. Μετά έχουμε τον Φιλίπ Φαντεμέρς, που είναι από την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικοδομών είσαστε και επαγγελματία του κλάδου και ξέρετε πολύ καλά τι θέλουν οι δημόσιες αρχές, οπότε πολύ χρήσιμη απόψή σας. Και τέλος από την Γερμανία έχουμε τον Έρμαν Πότς, έτσι. Ωραία. Με τη σειρά να πάρετε το λόγο λοιπόν. Πέντε λεπτά ο καθένας, έχουμε και διαφάνειες. Οπότε, η γραμματεία εδώ θα κρατάει το χρονόμετρο. Ρόμπερτ Χάν λοιπόν είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Κοιτάξτε, δεν έχω συνηθίσει να έρχομαι εδώ, ίσως κάνω λάθη. Εκπροσωπώ την σήμερα το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών για να σας βοηθήσω στην έρευνά σας για τις, για τις προκλήσεις όσον αφορά τις δημοσίες προμήθειες και καλύτερη τη θέσπιση νομοθεσιών και κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλεί το κενό με ερωτηματικό. Είμαι δικηγόρος και είμαι υπεύθυνο για τις εταιρικές σχέσεις, νομικές υπηρεσίες για τις ε, εταιρικές σχέσεις. Ανήκουμε στην Ένωση για την τοπική αυτοδιοίκηση της Βρετανίας και θέλουμε να επικουρούμε τους δημοσιοφορείς, όποιοι είναι αυτοί στην Αγγλία, ε, να προμηθευτούν τα πιο περίπλοκα προγράμματα που κυρίω μέσω των διαδικασιών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου γίνονται αυτέ οι διαδικασίε. Προαναφέρθηκε. Μακάρι να μπορούσα να έρθω εδώ με μια ρόδινη άποψη, αλυσορροπημένη άποψη, αλλά έχω μόνο ένα πεντάλεπτο και δεν έχω αυτή τη δυνατότητα κάθε μέρα, οπότε θα σα δώσω του κακού τίτλου και λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα ε, εν είδη προημίου να θέσω το πλαίσιο. Όλοι θα γνωρίζετε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ενδεχομένω μοναδικέ οικονομικέ περιστάσει και αυτό οδήγησε ε, σε τραπεζική κρίση και χρηματοδοτήσεω όχι μόνο στον ΕΒ και αλλού έχουμε ύφεση και πολλέ επιχειρήσει χρεοκοπούν. Υπάρχει μια πραγματική πρόκληση μπροστά μα. Ταυτόχρονα λυπάμαι να πω ότι η εμπειρία μου είναι ότι οι διαδικασίε προμηθειών που θα έπρεπε να βοηθούν τον ανταγωνισμό να βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται έχουν γίνει πιο δαπανηρές, πιο περίπλοκες και πράγματι αμφισβητούμενες νομικά για πολλούς που αναμειγνύουν τη διαδικασία. Ε, υπάρχει μια ε, κουλτούρα προσφυγής, υπάρχει αμφισβήτηση νομολογίας του δικαστηριού και θέματα που αφορούν τον περίπλοκο χαρακτήρα των διαδικασιών που επηρεάζουν τις αρμοδίου φορεί και εκείνου που βάλουν προσφορέ. Ε, επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Θα ήθελα απλώ να αναφερθώ σε ένα-δύο θέματα. Ετοιμάσαμε ένα έγγραφο το οποίο σα υποβάλαμε, όπου αυτά τα θέματα αναφέρονται λεπτομερώ. Θα ήθελα καταρχά να πω εκ νέου από την ταπεινή έποψη αυτού που ασχολείται στην πράξη με αυτά τα θέματα, βλέπουμε πολλά ζητήματα που τίθενται χωρί να υπάρχει σωστό συντονισμό. Αυτό αισθανόμαστε. Κάποιε από τι πρωτοβουλίε αναφέρονται σε ήπια μέτρα και νομοθετικά μέτρα. Είναι δύσκολο να δούμε αν υπάρχει ιεράρχηση και πού εντάσσονται όλα τα μέτρα σε όλο το τοπίο τη ε, και αυτό προσθέτει στη γενικότερη σύγχυση που επικρατεί. Επόμενη διαφάνεια. Ταυτόχρονα έχουμε μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τη θεμελιώδη αρχή που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι αυτή η αρχή. Ότι η τοπική φορή, η τοπική αυτοδιοίκηση, οποιοδήποτε δημόσιο φορέ, περιφερειακό ή τοπικό, θα πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιο κατά πόσο θα πρέπει μια δραστηριότητα θα διατεθεί στην αγορά ή όχι για ανταγωνισμό. Ε, ελπίζουμε αυτή η θεμελιώδης αρχή να γίνεται σεβαστή, να έχει ότι έχει διαβρωθεί ε, και θα θέλαμε να ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής συνθήκης της Αβώνα. Τώρα για να πάμε στο ψητό της παρουσίασής μου. Οι νέες διαδικασίες, διοικητικό κόστος στα πλαίσια της όλης νοοτροπής που έχει δημιουργηθεί. Και εδώ βρένει και το ερωτηματικό για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά πόσο καλύπτει το κενό. Λοιπόν, σαν νομικός θα έλεγα ότι είναι σωστό και δίκιο και είναι αρμόδιε φορέ στο δικαστήριο, να ερμηνεύει την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να απαντά σε ερωτήματα που δημιουργούνται κατά την πρακτική εφαρμογή του νόμου όσον αφορά τι προμήθειε. Όμω, κάποια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δημιουργεί ε, σύγχυση και του τελευταίου μήνε. Ε, έχει, μπαίνει σε, σε νέα χωράφια ο νόμος για την προμήθεια και έχουμε διάφορες υποθέσεις που έχουν προκύψει και λήφθησαν αποφάσει. Και αποφάσει που ελήφθησαν σε κάποιε περιστάσει έχουν απροσδόκητε συνέπειε, αρνητικέ συνέπειε. Για να σα δώσω και κάποια παραδείγματα. Στον τομέα μου. Ανταγωνιστικό διάλογο και περίπλοκα προγράμματα, σημαντικά προγράμματα και έργα. 9 με 18 μήνε χρειάζονται από τη διαδικασία επιλογή μέχρι, μέχρι το στάδιο τη ανάθεση. Μέχρι να αντιμετωπιστούν τα διάφορα εμπορικά και οικονομικά θέματα και μας λέει η νομολογία του δικαστηρίου που επήλθε σε πλαίσια, είναι πολύ δυσ... Ε, ταχεία διαδικασία, ότι πρέπει να έχουμε κριτήρια να κάνουμε σταθμίσει. Όλοι οι νόμοι είναι αμετάβλητοι. Δεν πρέπει να ρυθμίζουμε τι λεπτομέρειε για να ταιριάξουμε στην αγορά. Και τι είχαμε σε 18 μήνε. Από εικόνα φτάσαμε σε ανησυχητική εικόνα. Και οι αρχέ πρέπει να είναι ρεαλιστικέ. Πρέπει να αντιδρούν επί τόπου και δυστυχώς επειδή υπάρχει αυτή η αμφιβολία όσον αφορά τον νόμο, εμφισβήτηση του νόμου και κατά πόσο είναι αποτελεσματικό ο νόμο, αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Και μάλιστα μια εποχή που ο ανταγωνιστικό διάλογο ε, προχωρούσε μια χαρά και βλέπαμε κάποια ωφέλη. Στο τέλο τη διαδικασία τώρα έχουμε σημαντικό πρόβλημα με του χρηματοδότε που δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα στον συναλλαγή, γιατί φοβούνται μην τα χάσουν αν υπάρξει προσφυγή και η συναλλαγή θεωρηθεί άκυρη για κάποιο λόγο. Μα λένε ότι δεν μπορούμε να επανεξετάσουμε αυτά που ήδη έχουν εξεταστεί σε, πρώιμο στάδιο επιλογής. Είναι λογικό να μην επαναξεταστούν οι οικονομικές συνθήκες ε, που διέπουν τον φορέα στον οποίο θα κάνει την ανάθεση και θα είναι τέλο σου για τα επόμενα 30 χρόνια. Εγώ θα λέγω ότι είναι λογικό να μπορούμε να επανεξετάσουμε τα στοιχεία. Λοιπόν, συμπεράσματα, πώ πετάει ο χρόνο όταν μιλάει κανεί. Καλωσορίζουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να συμμετάσχουμε πλήρω στην αναθεώρηση των οδηγιών για τι δημόσιε προμήθειε, όταν αυτό συμβεί, παροτρύνουμε θεσμικά όλα τη Ευρωπαϊκή Ενώση να λάβουν υπόψη την, την ε, εμπειρία αυτών που εφαρμόζουν τον νόμο στην πράξη. Θέλουμε αξία. Αυτό είναι ο νόμο ε, των κρατικών αυτών των προμηθειών. Δεν είναι να αποφεύγουμε τι επιθέσει κάποιων που αφισβητούν κατά πόσο έγινε σωστά η ανάθεση. Θέλουμε να παρέχονται ε, υπηρεσίε σωστά. Αυτό ο σκοπό. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσει μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει Νομίζω ότι άξιζαν τον κόπο τα λεφτά που μιλήσατε. Εμείς οι πολιτικοί θέλουμε να ακούμε την ομοία αλήθεια. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στον καθηγητή Ροντρίγκε, που θα μας δώσει την ακαδημαϊκή οπτική γωνία του θέματος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, δεν θα σας παρουσιάσω την άποψη κάποιου οργανισμού, κάποιου φορέα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται περισσότερο αντικειμενικός. Γιατί θέλουμε να εξελιχθεί το πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ερώτημα που θα προσπαθήσω να απαντήσω πριν περάσω στο πώς να το αλλάξουμε. Ε, λοιπόν, υπάρχει ένα πλαίσιο. Επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ως εξή. Ότι υπάρχει μια αίσθηση δυσαρέσκειας από την τοπική αυτοδίκηση εδώ και αρκετά χρόνια που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Και δεν μπορείτε εσείς να γνωρίσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά αποτελεί και ένα άλοθη για να αλλάξουν τα πράγματα και το είπατε κι εσείς στην αρχή. Από την άλλη μεριά έχουμε και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δίνει κάποια δείγματα εξελίξεων. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να πάρουμε το τρένο, τώρα πρέπει να βγούμε στο τρένο. Συνεπώς, δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, πώς θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα στο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων και δεύτερον πώς θα παγιώσουμε μέσα στις υπάρχουσες οδηγίες τις εξελίξεις εξαιτία της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, τι είναι οι συμβάσεις παραχώρησης. Για να μπούμε λίγο και στα πιο τεχνικά στοιχεία, υπάρχει μια διαφορά Όσον αφορά τον ορισμό, πρέπει να τον γνωρίσουμε αυτό, ανάμεσα σε αυτά που λέει οι οδηγίες για τον ορισμό της παραχώρησης και σε αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ορίσει την παραχώρηση. Πρόκειται για το κριτήριο του κινδύνου, το οποίο είναι περισσότερο παρόν στην ομολογία του δικαστηρίου από ότι στον ορισμό που έχουμε στα κείμενα των οδηγιών. Συνεπώ, μια από τι πρώτε εξελίξει που πρέπει να κυνηγήσουμε είναι να είναι περισσότερο συμβατά τα κείμενα μεταξύ του, τα κείμενα με την ομολογία. Οι οδηγίε με την ομολογία. Δηλαδή, να διευκρινίζεται η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους συμβάσεων, παραχώρησης, με μια αυτόνομη ίσως οδηγία. Και δεν πρέπει να αποφεληθούμε από την ανακοίνωση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συμπράξει ιδιωτικού δημοσίου τομέα, όπου λέει ότι θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευση για να σκεφτεί μήπως πρέπει να υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Να λοιπόν μια ευκαιρία την οποία πρέπει να δράξουμε δίχως άλλο, σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο σκέλος πρέπει να δώσουμε περισσότερη ευελιξία, ελαστικότητα στις τοπικές δικήσεις για να ε, χειριστούν τις υπηρεσίες τους. Και γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο εύρος ε, ρεαλισμού που συνοψίζεται πάρα πολύ καλά στην τελευταία απόφαση CSRL που σας συστήνω να διαβάσετε, γιατί όντως βλέπετε όλες τις περιπτώσεις των τελευταίων ετών. Επιμένω επίσης και σε κάτι άλλο, στην αμοιβαιότητα και στην ε, διακοινωτική συνεργασία. Είχαμε την απόφαση της Κομισιόν κατά της Γερμανίας, με μία εξαίρεση όμως υπέρ της διακοινωτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή την εξέλιξη πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στα κείμενα για να παγιωθεί. Γιατί αυτά που λέει το δικαστήριο μια μέρα μπορεί να τα πει αλλιώ μια άλλη μέρα. Τέλος, να διασφαλίσουμε προκειμένου να ευνοηθούν οι διαδικασίες σύμπραξης ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Και εδώ υπάρχει κάτι θετικό. Στην περίπτωση εταιριών μικτής οικονομίας, ΑΚΟΣΕΤ, πέρυσι, εκεί είχαμε μια απόφαση όπου το δικαστήριο μιλάει για ευελιξία, για ρεαλισμό υπέρ τέτοιων επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει να πάρουμε το τρένο έγκαιρα, να ξεκινήσουμε έγκαιρα και εν κατακλείδη. Πρώτα απ' όλα, ε, μιλήσαμε για ερμηνευτική ανακοίνωση. Όντω θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη. Θα μπορούσαμε όμω να σκεφτούμε και άλλε λύσει. Μια οδηγία για τι συμβάσει παραχώρηση. Όμω αυτό το οποίο μετράει είναι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη διάρθρωση των εξελίξεων στην ομολογία και ε, των μέσων που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας για τις δημόσιες συμβάσει. Γιατί εδώ υπάρχει μια σχέση. Ο ρεαλισμό του δικαστηρίου γίνεται για καλύτερη οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών. Συνεπώ πρέπει να υποφεληθούμε από αυτέ τι εξελίξει και από το ρεαλισμό στι δημόσιε αγορέ για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ για τόσα μα είπατε. Πραγματικά όπως φαντάζεστε, ως Βρετανός πολιτικός που είμαι, εσείς μιλάτε για ευελιξία και ρεαλισμό. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν νομίζω τους Βρετανούς. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωραία. Πώς θα καταλήξουμε σε νομική βεβαιότητα με αυτή την ελαστικότητα ε, και τον πραγματισμό δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο κύριος Φαντεμέρς τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Φαντεμέρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ομοσπονδία η Ευρωπαϊκή του Κλάδου Οικοδομών αποτελείται από 34 ομοσπονδίες μέλη, από 29 χώρες και συμπεραβάνονται εκεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα των οικοδομών και των πολιτικών μηχανικών. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι οι Οδηγία του 2004 ε, είναι καλές, αρκούν και είναι καλά προσαρμοσμένες στην τρέχουσα κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Εμείς επιμένουμε λοιπόν ότι πρέπει να τηρούμε τη συνθήκη. Σωστή εφαρμογή των αρχών της, ε, θεμητός ανταγωνισμός, διαφάνεια, ίση μεταχείριση κλπ. κλπ. Συνεπώ, οι κατευθυντήριε γραμμέ και άλλα ερμηνευτικά κείμενα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν αποτελούν δεσμευτικά νομικά κείμενα. Οι γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα έκαναν να συντονιστούν καλύτερα μεταξύ του για να υπάρχει συνοχή στι οδηγίε του. Επί του παρόντο, η νομοθεσία για τι δημόσιε αγορέ χρειάζεται σταθερότητα προκειμένου να υπάρξει περισσότερη νομική ασφάλεια για του εμπλεκόμενου. Εξάλλου θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δώσει επικοδομητικέ απαντήσει όσον αφορά τι αβεβαιότητε που αντιμετωπίσαμε στην πράξη η συνεργασία δημοσίου-δημοσίου τομέα, έτσι όπω έχει εξελιχθεί, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει παράλληλε αγορέ οι οποίε να ξεφεύγουν από του κανόνε των δημοσίων αγορών και να αποκλείουν του ιδιωτικού εταίρους. Πρόκειται για αγορέ που δεν είναι δημόσιε. Στον τομέα των, συμπράξεων, των θεσμοποιημένων συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου τομέα, ε, έχει προσφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αρκετέ αποσαφηνήσει, οπότε δεν χρειάζονται επιπλέον διαδικασίε. Στον τομέα τώρα τη παραχώρηση υπηρεσιών, η τήρηση των συνθηκών είναι κάτι αναγκαίο, αλλά και φτάνει από μόνο του. Δεν χρειάζεται λοιπόν ειδική νομοθετική ρύθμιση. Αν παρόλα αυτά προβλέπετε κάτι τέτοιο, το πιο λογικό θα ήταν να επεκτείνουμε του κανόνε που ισχύουν για την παραχώρηση ε, έργου και στην παραχώρηση υπηρεσιών διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα τα οποία απαντώνται σήμερα έχουν να κάνουν περισσότερο με τη μεταφορά του δικαίου του ευρωπαϊκού στο εθνικό δίκαιο ή οφείλονται σε κακή πρακτική, κακή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αν παρόλα αυτό χρειάζεται μια αλλαγή στις υπάρχουσες οδηγίες, τότε πρέπει να προσέξουμε να υπάρξει συνοχή με τις άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις. Να αποφύγουμε νέα ερμηνευτικά κείμενα, να μην δημιουργήσουμε νέα προβλήματα, νέα κενά και να φροντίσουμε για την πρόθεση της καινοτομίας στις δημόσιες αγορές. Το θέμα της καινοτομίας είναι πάρα πολύ σημαντικό στις δημόσιες αγορές και μπορεί να γίνει μόνο εάν επιλέγουμε συστηματικά τις ε, πιο αποδοτικές οικονομικά λύσεις. Να λάβουμε υπόψη μας και τον κύκλο ζωής του κτηρίου και της υποδομής. Οι αναλλακτικές λύσεις από μια επιχείρηση Εφόσον δεν απαγορεύονται, μπορούν να επιτρέπονται, αλλά μόνο σε θελοντική βάση. Τέλος, το απόρριτο των προσφορών θα πρέπει να τηρείται απόλυτα, γιατί δεν είναι δυνατόν ιδέες καινοτόμε να κλέβονται εντό αγωγικών και να ανακυκλώνονται σε νέες προσφορές. Τέλο, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σα και σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που είναι οι επιχειρήσει εντό αγωγικών τρίτων χωρών που έχουν πρόσβαση στι δημόσιε ευρωπαϊκέ αγορέ. Τέτοιε επιχειρήσει δεν έχουν του ίδιου περιορισμού όπω έχουν ιδιωτικέ επιχειρήσει όσον αφορά τον κίνδυνο ή το κόστο. Είναι απαράδεκτο να επιτρέπονται τέτοιε πρακτικέ στην εσωτερική αγορά, ιδιαίτερα για projects τα οποία χρηματοδοτούνται και από, την, από ευρωπαϊκά χρήματα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρειάζεται επίση να τηρούν τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ και για κοινωνικού παράγοντε και για περιβαλλοντικού παράγοντε, όπω σέβονται και οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίε που κάνουν μεγάλες οικονομικές προσπάθειες για να ε, μας παρουσιάσουν προσφορές που να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Επίσης, όταν έχουμε κατά 30% χαμηλότερες τιμές δεν μπορεί να τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεπώς πρέπει οι αρχές να εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια τέτοιες αρχές και να βλέπονται αν δικαιολογείται η χαμηλή προσφορά που κάνουν. Αν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λοιπόν ε, θέλουμε να έχει μία ε, εσωτερική αγορά ανοιχτή πρέπει και να την προστατεύει κατά του dumping του κοινωνικού ή του περιβαλλοντικού. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία ή να περιοριστούμε να αποτελούμε το καλό παράδειγμα. Η Ομοσπονδία μας είναι πεπισμένη για το ότι η αρχή της αμεβαιότητας πρέπει να τηρείται αυστηρά. Στην αντίθετη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποβάλει τις επιχειρήσεις από τρίτες χώρες στις ίδιες συνθήκες που προβλέπονται και για τις ευρωπαϊκές. Δηλαδή να υπάρχουν στοχοθετημένοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ε, αγορών από τέτοιες επιχειρήσεις. Η Ομοσπονδία μας ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια τις διάφορες πτυχές αυτής της υπόθεσης η Ομοσπονδία μα και οι εταίροι μα, οι σε επίπεδο, θέλουν με την εμπειρία του να βοηθήσουν για την καλύτερη δυνατολάση. Τα πέντε λεφτά που μου δώσατε είναι λίγα. Ε, ξεπέρασα το χρόνο μου, το ξέρω, αλλά η επιχειρηματολογία μα με περισσότερε λεπτομέρειε βρίσκεται στο τραπέζι με τα διάφορα έγγραφα και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσει έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαντεμέσ. Ξέρω ότι η κυρία και ιδιαίτερα άκουσε την τελευταία σας παρατήρηση. Θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει αργότερα, διότι έχουμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι σημαντική για το θέμα αυτό. Και τέλος, ε, στο τμήμα αυτό να δώσω το λόγο στον Νόρμπερτ Πότς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, ευχαριστώ ε, την κυρία Ρούλε για την δυνατότητα να μιλήσω εδώ σήμερα. Εκπροσωπώ σήμερα 13.000 ε, ε, φορείς της, ε, τοπικούς φορείς της Γερμανίας και τα τρία και τα τρία επίπεδα του δημοσίου στην Ευρώπη, ομοσπονδιακό, σε και τοπικό επίπεδο, ε, ε, αναθέτουν κάθε χρόνο ε, έργα 260 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου, φιλική διαδικασία για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ σωστά η κυρία Ρίλε είπε ότι αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, η οικονομική κρίση αλλά και η νέα νομική βάση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας αποτελούν νέα δεδομένα και κατά τη γνώμη μας θα πρέπει η αποδοχή του, δικαίου που διέπει τι δημόσιες συμβάσεις να βελτιωθεί Θέλω να σας ε, αναφέρω τους τομείς όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Ε, καταρχήν, ο προσανατολισμός του δικαίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, να σέβεται το, τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επικουρικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ε, θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε περισσότερη πρακτική ε, βοήθεια. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι το δίκαιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις ε, δεν ε, θα πρέπει να διέπεται από αναλογικότητα και ε, σίγουρα μπορεί να συζητήσει κανείς ε, σχετικά με τους δικαιολογημένους στόχους, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να μπορούν να εξεταστούν από τους Δήμους. Ισχύει δηλαδή και εδώ η αρχή της αναλογικότητας. Το λιγότερο μερικές φορές είναι περισσότερο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ευρύτερο περιθώριο ευελιξίας και από τις πλευράς των υποψηφίων και από πλευράς της αναθέτουσας αρχής. Ε, με ανοιχτές διαδικασίες η δυνατότητα ε, διαπραγματεύσεων ε, μπορεί να διευρυνθεί. Επίσης Υπάρχει δυνατότητα να απλοποιηθεί η διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, ενισχυμένη δυνατότητα για τους ε, υποψηφίους να επιλέγονται, ε, να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή. Και πέμπτο, ασφάλεια δικαίου. Βλέπουμε ότι στην διαδικασία σημειώνονται πολλές παραβιάσεις οι οποίες δεν ε, ε, ε, τιμωρούνται επαρκώς. Πολύ συγκεκριμένα, δημοτική συνεργασία. Να αναφερθώ στις τρεις μορφές συνεργασίας, κοινοπραξίες δημοσίου-δημοσίου. Κατά τη γνώμη μας, αυτός είναι αυξανόμενος, ε, αναπτυσσόμενος τομέας για το μέλλον. Να σας αναφέρω για παράδειγμα την παροχή ε, ύδατος. Ε, είναι όμως και ένα θέμα το οποίο συνδέεται στενά με την επικουρικότητα στην απόφαση της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη Στατράνικουν Χάμπουργκ. Ε, δεν δίδονται ε, ε, εντολές σχετικά με την... Δεν υπάρχει απαγόρευση συνεργασίας μεταξύ Δήμων αρκεί να μην υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή για να μην εμπίπτουν στους κανόνες δημοσίων συμβάσεων. Όσον αφορά τις κοινοπραξίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ε, το ε, ΔΕΚ έχει επίσης ε, διευκρινίσει την κατάσταση. Θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται το δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων. Δεν είναι απαραίτητη ο διπλός διαγωνισμός και η δυνατότητα και ε, η δυνατότητα ε, ανοίγματος κεφαλαίου ε, μιας δημόσιας επιχείρησης δεν οδηγεί αυτόματα σε εφαρμογή του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων. Και τέλος έχουμε τις συμβάσεις παραχώρησης. Εδώ θέλουμε διαφάνεια, ανταγωνισμό και ίση μεταχείριση οι κοινοτικές ενώσεις, οι δημοτικές ενώσεις της Γερμανίας ε, θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελικτία και για τα συγκεκριμένα θέματα τη της κοινοπραξίας ιδιωτικού δικαίου, ε, της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων ε, φορέων και στις συμβάσεις παραχώρησης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν θέλουμε πάντως πρόσθετες νομοθετικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. πολύ σαφή αυτά που μας είπατε. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο χρόνο τώρα για σχόλια από πλευράς μελών και αν έχουμε χρόνο θα επανέλθω, θα δούμε πώς θα τα πάμε. Καταρχάς, θα ζητήσω από την Χάιντι Ρούλε, την εισηγήτριά μας, αν θέλει να θέσει κάποια ζητήματα στους εμπειρογνώμονες και μετά έχουμε κατάλογο ομιλητών που ετοιμάζουμε. Ας ακούσουμε πρώτα τους ε, σκιώδεις και μετά μιλάω, λέει η κυρία Ρούλε. Διότι είχα ήδη την δυνατότητα να εκφραστώ. Πολύ γενναιόδορη, λέει ο πρόεδρος, κύριο Σφάμπ. Κύριο Σφάμπ Βάιλε Στάλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, λέω στα αγγλικά, αλλά τώρα θα συνεχίσω στα γερμανικά. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρούιλε, καταρχήν ε, βρίσκω πολύ ε, ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της συζήτησης ως συντονιστές ε, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ε, επιλέξαμε για την αρχή της θητείας μας την ακρόαση αυτή για να εξετάσουμε εγκαίρως όλες τις πτυχές του δικαίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τα ε, συμφέροντα των ε, Δήμων και των τοπικών ε, αρχών, των αναθέτουσων αρχών. Να στραφώ πρώτα στον εκπρόσωπο της ΦΙΕΚ. Με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί Δημοσίων Συμβάσεων φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, δεν είναι αρκετά προστατευμένες κατά του αθέμητου ανταγωνισμού. Ε, φοβάμαι ότι με την απόφαση που αφορά τον, ε, την κάτω σαξονία και ρωτώ, μου φαίνεται ότι η απόφαση αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα ούτε των επιχειρήσεων ούτε των αναθετουσών αρχών. Στον τομέα των οικοδομών ε, στη Γερμανία, στη χώρα μου, υπάρχει ε, βασικός μισθός, ελάχιστος μισθός και εάν επιτρέψουμε υπερβολική ελευθερία ε, στη, στα κράτη-μέλη ε, με τους διαφορετικούς βασικούς μισθούς που ισχύουν στην κάθε χώρα ε, δεν θα είναι εύκολο να έχουμε μια καλή λύση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κύριε Πότσε, μιλήσατε για αποδοχή του δικαίου που διατηρεί τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη και ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποδοχή αυτή υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες ε, που αφορούν τις ε, τους μικρούς δήμους που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την γνώση των κανόνων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Ε, να ξεκινήσω από τον κύριο Πόλτς. Η συζήτηση μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι από τη μία μεριά στη Γερμανία και σε άλλα κράτη-μέλη ε, υπάρχει επιθυμία για περισσότερη ευελιξία. Από την άλλη ακούω από τους ανθρώπους ότι θέλουν περισσότερη ασφάλεια δικαίου αυστηρούς κανόνες ε, σύμφωνα με τους οποίους να μπορεί να προσανατολίζεται κανείς. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Μήπως ε, μπορείτε να μου πείτε τι βρίσκεται πιο σημαντικό, ειδικά για τους μικρούς δήμους που θα πρέπει να ε, δημιουργήσουν ανάπτυξη ε, στην περιοχή τους. Αναφέρθηκε και το dumping από τις τρίτες ε, χώρες. Αυτό το ανέφερε ο κύριος από τον τομέα των οικοδομών. Αυτό ισχύει όμως και για σας και για τις άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή συνάπτουμε συμβάσεις με τρίτες χώρες, συμβάσεις γειτονίας. Το Κοινοβούλιο συμμετέχει στις ε, συμβάσεις αυτές ε, με μέσω της ε, Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Εννοείτε τις χώρες εσείς με τις οποίες ήδη έχουμε τέτοιες συμβάσεις ή εννοείτε τις άλλες γειτονικέ μας χώρες, την Ουκρανία και άλλες. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για την περαιτέρω εργασία μας. Επίσης κύριε Πόρτς, μιλήσατε για έλεγχο των κριτηρίων. Αυτό βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτός ο έλεγχος των κριτηρίων και τα κριτήρια που εσείς φαντάζεστε ε, ε, μιλάτε για παράδειγμα για ε, τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές για ένα πολύ καλό και χρήσιμο ξεκίνημα στην ακρόασή Να στραφώ στον συνάδελφο Βασάκ που μίλησε για κανόνες δημοσίων συμβάσεων. Βρίσκω ότι είναι εξαιρετική η ιδέα σας, αν και αυτή τη στιγμή πολλές τοπικές αρχές για λόγους περιορισμών στον προϋπολογισμό. Εγώ προέρχομαι από τη Σκωτία και εκεί ισχύει αυτό. Πολλοί μιλάνε για ε, εκπαίδευση. Άκουσα για παράδειγμα ότι έχουν γίνει περικοπές ε, στην, εκπαίδευση, στη γλωσσική εκπαίδευση δασκάλων στα δημοτικά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αλλά εάν ε, κόβουμε τις δαπάνες σε τέτοια, αν περικόπτουμε τις δαπάνες σε τέτοιους τομείς, πώς θα περάσουμε τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να Επιμείνουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, ομιλητές. Ε, ε, Βρίσκω υποποίηση για το άρθρο 19 από λομπίστες, από ομάδες συμφερόντων και Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να προωθήσουν ιδιαίτερα τους, τομείς, τους κανόνες αυτούς. Έχει να κάνει με την πρόσληψη από δήμους ε, ατόμων με αναπηρία. Λένε όμως ότι δεν γίνονται αρκετά στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τους συλλογισμούς σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω προ το τελευταίο θέμα, νομίζω ότι θα καλυφθεί στο δεύτερο μέρος τη ακρόαση και όχι στο πρώτο. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να είναι σύντομοι με τι ερωτήσει του, διότι θα ήθελα οι εμπειρογνώμονε να προλάβουν να απαντήσουν. Ε, Έγκελ Γκέπχαρτ και η κυρία Φερχέν νομίζω από την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και η κυρία Ρούιλε. Ε, παρακαλώ, κυρία Έγγελ. Ευχαριστώ. Θα απευθυνθώ προς τον καθηγητή Ροτρίγκε περισσότερο. Στο βαθμό που φαίνεται να αποκριστάλλωσε ότι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε απαραίτητα περισσότερη νομοθεσία, τουλάχιστον όχι σε μαζικό επίπεδο, όλοι θέλουμε να έχουμε πρακτική εφαρμογή των ισιών κανόνων. Αναφερθήκατε στη δυνατότητα ξεχωριστής οδηγίας ένα πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις ε, κορίσεις όπως είπατε και δεύτερον για τη σύμπραξη δημοσιο ιδιωτικού τομέα και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά που θέτουμε ε, διαφέρουμε καταρχήν επ' αυτού και αν ναι, θα εκτιμούσα κάποιες λεπτομέρειες επ' αυτού και σίγουρα θα είσαστε σε θέση να μας δώσετε αυτές τις λεπτομέρειες ε, διευκρινήσεις. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ σε μια αντίφαση που άκουσα από τον κύριο Ροντρίκες, τον οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Ε, και σε αυτά που είπε ο κύριος Πόρτς. Ο κύριος Πόρτς είπε ότι θα πρέπει να αφήσουμε την νομοθεσία ως έχει, να μην κάνουμε καμία τροποποίηση. Ενώ ο κύριος Ροτρίκες ε, συμβούλεψε τις ε, αρχές που ε, μπορεί να εξάγει κανείς από τα, τις αποφάσεις του ΔΕΚ θα πρέπει να τις ε, εισάγουμε στο δίκαιο για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου διότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σίγουροι ότι τα δικαστήρια θα, θα παραμείνουν σε αυτά που έχουν αποφασίσει στο παρελθόν. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση κύριε Ροντρίγκε και κύριε Πόρτς. Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα. Θα ήθελα περισσότερες εξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολλοί από μας είχαμε την απορία αυτή. Ευχαριστώ που το διευκρινίσατε. Κύριε Βαχιάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, διαπιστώνω ότι και από την δημοτική πλευρά αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων ε, δεν ε, Υπάρχει απαραίτητα επιθυμία για νέα νομοθεσία, αλλά καταρχήν περισσότερη διαφάνεια, παρουσίαση, ερμηνεία, ε, όπως για παράδειγμα έχουμε το τελευταίο καιρό μέσα από το ΔΕΚ ε, και κυρίως για τους Δήμους μεγαλύτερη διαφάνεια στην παρουσίαση και στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη ε, να διεξάγονται καλύτερα οι διαδικασίες ε, που έχουν να κάνουν με την ανάθεση ευρωπαϊκών έργων. Ε, οι γενικές διευθύνσεις ίσως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν φτάνει μία μέρα για τους Δήμους για να αφομοιώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Πώς φαντάζεστε εσείς να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία αυτή, να μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίλε. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ερωτήσω τον κύριο Χέν που έχει ε, πρακτική εμπειρία στον τομέα του ανταγωνιστικού διαλόγου. Πιστεύω ότι ο ανταγωνιστικός διάλογος αποτελεί κεντρικό σημείο. Υπόθηκε ότι ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να ε, αρκεί για να γίνουν πιο ευέλικτες ε, οι συμβάσεις παραχώρησης. Και μια ερώτηση προς τον κύριο Ροντρίκες που έχει να κάνει με το θέμα της νομοθεσίας αυτό συνδέεται και με αυτό που είπε η κυρία Κέπχαρτ, αλλά θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Ε, έχω μιλήσει με πολλού ενδιαφερομένους στον τομέα αυτών, μεταξύ άλλων με το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, ε, που μου εξήγησαν ότι μια ρύθμιση για τις συμβάσει παραχώρησης ε, θα ήταν μόνο αποδεκτή εάν συνάδει με το γαλλικό μοντέλο. Αυτό το λέει εδώ και χρόνια, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και μήπω θεωρείτε κι εσεί ότι νομοθεσία στον τομέα της, ε, των συμβάσεων παραχώρησης θα σημάνει ε, στένεμα των περιθωρίων εντός των κρατών μελών, περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερο γραφειοκρατικό άχθος. Ίσως θα έπρεπε ως πρόεδρος και ως κοιόδης να προβώ και εγώ σε σύντομο σχόλιο. Με διέφερε η παρουσίαση του κ. Χάνς που αναφέρθηκε σε θεμελιώδη αναθεώρηση και αξιολόγηση των οδηγιών, αλλά όχι νέες οδηγίες. Κάποια από τα θέματα που όλοι θίξατε, νομίζω, αφορούν την πρακτική εφαρμογή περίπλοκης νομοθεσίας, επιτόπια εφαρμογή. Και επίση ότι οι πρόσφατες αποφάσεις και νομολογία ενεθάρρυναν από ό,τι φαίνεται πλέον ευέλικτη και πραγματιστική ερμηνεία. Το ερώτημα για μας ποιο είναι. Πρόκειται περί επιχειρησιακού θέματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο Ότως ώστε οι φορείς και οι κυβερνήσεις να αναθέτουσες αρχές κυβερνήσεις να συνεργαστούν. Ο θεσμικός μηχανισμός μετά, μέσω των οποίων λειτουργεί η κρατική προμήθεια σε διάφορες χώρες η σωστή προσέγγιση. Υπενθυμίζω ότι όταν πήγαμε στη Σουηδία πρόσφατα, η Επιτροπή μας, συναντήσαμε την αρχή ανταγωνισμού της Σουηδίας και μας ξεκαθάρισε αυτή η αρχή ότι είναι υπεύθυνη και για τις κρατικέ ε, κρατικές προμήθειες, διότι θεώρησαν ότι είναι θεμελιώδες θέμα για την ανταγωνιστική οικονομία. Θα ακούσουμε και τους Σουηδούς συναδέλφου σήμερα. Είπαν ότι υπάρχει ευστηρό έλεγχος Μήπως πρέπει να επιφορτήσουμε τις κυβερνήσεις με αυτό, να φροντίσουν για την πιο εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Αυτό είναι το ερώτημά μου τώρα. Φορώ το καπέλο του Προέδρου και καλώ τους τέσσερις από εσά, ξεκινώντας από τον κύριο Χαν και ακολουθώντα αντίστροφη σειρά, να μας δώσετε, αν μπορείτε, το ταχύτερο δυνατόν κάποιε απαντήσει Και πάντα μπορούμε να σα δώσουμε τη δυνατότητα να στείλετε κάποιο σημείωμα αργότερα. Ξεκινώντας το χρονόμετρο σας δίνω ένα λεπτό περίπου, είμαι και έτοιμος να είμαι ευέλικτος και μετά προχωρούμε στο επόμενο τμήμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω. Αν ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι τρόπος ευελιξίας, δεν σας δώσω τα καλά μαντάτα. Η διαπραγμάτευση και το στοιχείο του αγωνιστικού διαλόγου είναι κάτι θετικό, πάρα πολύ καλό κατά την απόψη μου ιδέα. Αυτοί που υποβάλλουν προσφορέ να μπουν σε μια αίθουσα και να δώσουν την καλύτερη λύση και να βοηθούν την καινοτομία είναι καλή. Είναι δαπανηρό το σύστημα και η κοινότητα των προσφορών αντιδρά. Μετά, η πρακτική εφαρμογή περίπλοκης νομοθεσία. Εάν υπήρχε ένας τρόπος, ο, ο ανταγωνιστικός διάλογος και όλη η διαδικασία στο τέλο κάπως να προσαρμόζεται, διότι εδώ δημιουργούνται τα προβλήματα στο τέλο. Όταν αυτοί που κάνουν, υποβάλλουν τις προσφορές ε, βλέπουν να αυξάνεται το κόστος και μπορεί να κερδίσει μόνο ένας. Αυτός που χάνει έχει κάθε λόγο να μπλοκάρει τον αντίπαλό του όταν έχει ε, αναλάβει την, ε, το έργο. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι λογικό να το εξετάζει αυτός που υποβάλλει προσφορές. Να εξετάζει τις έρευνες κλπ. Ένας να εξετάζει το θέμα και να μην εμπλέκονται και οι σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε και τα κέρδη έρχονται πιο εύκολα μετά. Στο τέλο τη διαδικασία λοιπόν υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Κάποια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Καθηγητή Ροντρίγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τι δύο ερωτήσει. Εάν πρέπει να ομοθετήσουμε και ανέ ναι, πώ. Ίσως να μην υπήρξα αρκετά σαφής προηγουμένως. Λοιπόν, είχαμε, είχα παραθέσει κάποια πράγματα με ερωτηματικά στο τέλο. Υποθεθήστο ότι προσπαθούμε κάτι να κάνουμε, διότι υπάρχει και ένα πρώτο σενάριο, όλοι είναι ικανοποιημένοι, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει όμω και μπορούμε να πούμε πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακολουθεί ένα νέο μονοπάτι, Α το αφήσουμε λοιπόν μόνο του να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι και να τροφοδοτήσει την ευελιξία της συνεργασίας, την ευελιξία των εξαιρέσεων κλπ. Αυτή είναι μια πρώτη επιλογή. Δεύτερη δυνατότητα, αν αποφασίσετε να προχωρήσετε πιο πέρα. Προφανώς ε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά τα εργαλεία τα νομοθετικά, υπάρχει η δυνατότητα αναθεωρήσεως των ισχυόντων ε, ή ένα αυτόνομο κείμενο. Ας δούμε τι γίνεται για τις παραχωρήσεις. Ο νομοθέτης αποφάσισε να καθορίσει επιτέλους το 2004 αυτές τις παραχωρήσεις και βλέπουμε ότι το ΔΕΚ χρησιμοποιεί ένα κριτήριο διαφορετικό. Διαφορετικό, όχι τόσο τελείω διαφορετικό, αλλά πιο ακριβέ. Πολύ πιο ακριβέ όσον αφορά την μετακύριση του κινδύνου. Μήπω θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο ορισμό που χρησιμοποίησατε. Την πάση περιπτώσει, το δικαστήριο ε, σα δημιουργεί κάποια παζοκεφαλιά. Λοιπόν, μπορεί να αναθεωρήσετε τα ισχύοντα για να συμπεριλάβετε τι εξελίξει. Δεύτερη δυνατότητα. Ενδεχομένω να δώσετε περισσοτερες δεπτομέρειε, λεπτομέρειες, συνεργασία μεταξύ εξαιρέσει εξαιρέσεις in-house εντός του οίκου. Όλα αυτά δεν αφορούν τις δημόσιες προμήθειες, δεν χρειάζεται να ενταχθούν στην οδηγία, είναι κάτι συγκεκριμένο, ειδικό. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο, δεν ξέρω. Διαπιστώνω απλώς ότι είναι, έχουμε την Κοντιτέλ Μπραπάντ, υπόθεση Ταμπούργ στην Γερμανία. Δεν είναι γαλλική ιδιαιτερότητα αποκλειστικά. Υπάρχει ένας κίνδυνος να επιβάλλει μια χώρα το μοντέλο της, διότι υπάρχει ε, ένα, μια νομολογία πολύ ανεπτυγμένη. Αλλά σκεφτούμε αν μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό για όλους και για τα 27 κρατημέλη αυτή, αυτά τα μοντέλα. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα. Εγώ δεν θα προτείνω θαυματουργές λύσεις, αλλά σκεφτείτε πολύ καλά αυτή τη διαφορά που αρχίζει να δημιουργείται. Ε, και δεν είναι ο μόνος Διαφορά μεταξύ κρατικής προσέγγισης του νομοθέτη στα μάλλον ακαμψίας του νομοθέτη και ευελιξίας που επιθυμούν αυτοί που εφαρμόζουν την νομοθεσία επιτόπου. Λοιπόν, μπορείτε να διαλέξετε και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντόπισα τις ερωτήσεις που απευθυνόταν περισσότερο προς τη ΦΙΕΚ. Ε, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό που έχει υπόψη της η ΦΙΕΚ δεν είναι η απόφαση της κάτω Σαξονίας. Υπήρχε κοινωνική διάταξη που ήταν ιδιαίτερη εκεί. Αυτό που θέλαμε να καταγγείλουμε είναι το κοινωνικό dumping κάποιων, κρατών, κάποιων επιχειρήσεων κρατικών τρίτων χωρών, κρατικών επιχειρήσεων που καταφέρουν να κατακτήσουν αγορές, ακόμα και αγορές που παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ωφελούμενες εκφεύγοντες από το κριτήριο κέρδους που πρέπει να σεβαστούν οι επιχειρήσεις μας έρχονται και κερδίζουν αγορές στην Ευρώπη, μερίδιος της αγοράς, στην εσωτερική αγορά, με μη ανταγωνιστικές τιμές. Και πιστεύουμε, έχουμε την άποψη, ότι τέτοια πρόσβαση στην αγορά δεν μπορεί, δεν επιτρέπει να... Δεν σέβονται, χωρίς να σέβονται περιβαλλοντικούς κανόνες και άλλους κανόνες αποκτούν αυτά τα μερίδια της αγοράς. Και λυπούμε που κάποιες χώρες λησμονούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που, που αυτές συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις που προσφέρουν και σε επιστούμε, ε, εφιστούμε την προσοχή επ' αυτής της πραγματικότητας. Εγώ ξέρω μόνο τον τομέα των οικοδομών, εκεί έχω την ευαισθησία μου. Αλλά είναι αρκετά ανησυχητική αυτή η πραγματικότητα για τις μεγάλες αγορές όπου, όπου ε, γίνονται ανταγωνιστικές αυτές τις εταιρείες χωρίς να σέβονται όμως τα κριτήρια τα Ακούστε Ακούστηκε μια σειρά ερωτήσει, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ο κύριο Σβάμπ ε, ρώτησε σχετικά με την ε, αποδοχή. Ε, εγώ θα ευχόμουν οι Δήμοι όταν εφαρμόζουν το το δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών ε, να μην πρέπει κάθε φορά να προσλάβουν ακριβούς ε, δικηγόρους ε, διότι θα πρέπει να γίνει λίγο, λιγότερο γραφειοκρατική η διαδικασία και αυτή είναι απάντηση και προς την κυρία Βάιλερ όσον αφορά την ευελιξία. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά αυστηρή η διαδικασία και υπάρχει ο φόβος από τους Δήμους να κάνουν λάθη αναφέρθηκα στην ε, μεγαλύτερη ευελιξία και είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα προεπιλογής των υποψηφίων ε, χωρίς ε, να είναι επαχθής η διαδικασία. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ναι, κυρία Βάιλερ, έχετε δίκιο όσον αφορά τι ε, κοινωνικέ πτυχέ. Ε, ε, δεν υπάρχει αντίρρηση ω προ την εφαρμογή των βασικών μισθών, αλλά με όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει υπερβολικά γραφειοκρατική διαδικασία για την αναθέτουσα αρχή. Η κυρία Κέπχαρτ έθεσε ένα ερώτημα. Εγώ είπα μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξία ε, των αναθέτουσων αρχών όσον αφορά τους ε, πιο στενούς τομείς. Έχει γίνει σαφές ότι έχουμε δύο τομείς ε, που εξαιρούνται από το ε, δίκαιο περί ε, δημοσίων ε, συμβάσεων, οι συμβάσεις παραχώρησης και οι κοινοπραξίες σε δημοσίου-δημοσίου. Η κυρία Ρούλερ αναφέρθηκε και στις συμβάσεις παραχώρησης είναι τόσο πολύπλοκες που αν θέλουμε ε, ανταγωνισμό θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και όσον αφορά τις κοινοπραξίες ε, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα είναι σαφής η θέση μας ε, ότι οι δήμοι μπορούν κάλλιστα να εφαρμόσουν τους κανόνες δεν χρειάζεται πλέον νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Uh, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τέσσερις ε, επαΐοντές μας για τις σαφέστατες, χρησιμότατες τοποθετήσεις τους, παρουσιάσεις τους και έχετε στους κίτρινους φακέλους και γραπτά που μας έδωσαν και κείμενα που μας έδωσαν. Η κυρία Ρούλε που είναι σκιώδης και εγώ θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά, θα εξετάσουμε λεπτομέρειες. Ε, δεν διευκολύνεται το έργο μας γιατί ότι μας θέσατε και άλλα ζητήματα, όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και ελπίζω να μπορέσετε να μας βοηθήσετε αν χρειαστούμε υπεραιτέρω διευκρινήσεις. Ας στραφούμε τώρα στο δεύτερο τμήμα. Θέλουμε να εξετάσουμε την νομικές, τις συνέπειες της νομικής αβεβαιότητας όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές και περιβαλλοντικές πτυχές ε, των διαφόρων ε, διατάξεων και τις συνέπειες του υπείου ε, της ήπιας νομοθεσίας, που θα καλείτε. Θα ήθελα ξανά να παρουσιάσω τους ομιλητέ, τους βλέπω όλους εδώ, είναι πιο γνωστά τα ονόματά σα κάπως. Να σας παρουσιάσω και να σας καλέσω ξανά να πάρει το λόγο για πέντε λεπτά ο καθένας. Η κυρία... Α, είναι μέλος της Business Europe και πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τις κρατικές προμήθειες από την Ορβηγία. Είναι, α, είναι νομικός. Σας καλωσορίζουμε. Η Νορβηγία είναι μέλος της εσωτερικής αγοράς και εφαρμόζει τις οδηγίες για κρατικές προμήθειες και φορά το λησμονούμε εδώ, οπότε είσαστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι εδώ. Πίτερ Νόρστατ μετά, από το Σουηδικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη κάποιων σημαντικότατων προγραμμάτων στη Σουηδία για την πράσινη προμήθεια. Μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε σήμερα τι έχετε να μας πείτε, όχι σε πολλές λεπτομέρειες, ίσως να μας ξυπνήσετε το ενδιαφέρον. Σχετικά με τα τεκτενόμενα στη Σουηδία, ανέφερα και τη Σουηδία προηγουμένως για τη γενική δουλειά που έχει κάνει για τις κρατικές προμήθειες και τον Κένεθ Κλάρκα, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων, στην Ομοσπονδία ε, ενώσεων υπηρεσιών, 800 ε, τέτοιε ενώσει εκπροσωπεί η κυρία αυτή μάλλον, και είναι επικεφαλή τη μονάδα πολιτική που συμπεριλαμβάνει την ευθύνη για τι ε, δημόσιε προμήθειε και τη συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τον κύριο Γκεγιόνγκ που εκπροσωπεί τη όμως Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιτροπιών Διασύνδεση για την Κοινωνική Στέγαση άλλη μια α, πτυχή όσον αφορά τις κρατικέ κρατικές αυτές προμήθειες. Η κυρία Γιούνες λοιπόν έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την θερμή σας υποδοχή κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Η Business Europe θεωρεί ότι αρκούν οι ρυθμίσεις που έχουμε μέχρι τώρα για τις δημόσιες συμβάσεις. Υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός επίσης. Και αυτό είναι ο βασικός στόχος, νομίζω, προκειμένου να καταπολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Οι δύο οδηγίε που έχουμε δεν θα έπρεπε να δεχτούν πιέσεις. Νομίζω ότι η ενσωμάτωσή του στο εθνικό δίκαιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχουμε στην εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, που είναι πολύ βασικέ για την απασχόληση, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Επίση, χρειάζονται μέτρα, αλλά για πρακτικούς λόγους δεν θα πρέπει να είναι εξίσου εκτενείς όπως και όταν μιλάμε για πάνω από το όριο. Η πρόσβαση στι δημόσιε συμβάσει τώρα. Είναι οι αρχέ των δημοσίων συμβάσεων που πρέπει να φροντίσουν για πρακτικέ για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, να φροντίσουν να υπάρχει ενδεχομένω ε, ε, το έργο να κοπεί σε κομμάτια για να μπορούν να συμμετέχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, να γίνεται δημοσιοποίηση σε κεντρικέ ιστοσελίδε κλπ. Είναι πολύ βασική αυτή η δημοσιοποίηση και είναι πολύ βασική και η διαφάνεια. Η Business Europe πιστεύει ότι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δεν χρειάζονται. Σίγουρα υπάρχει θέμα κινδύνου και θέμα διάρκειας, πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εξελίξεις και στις συνθήκες. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ λεπτομερείς. Οι δημόσιες συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν εργαλείο για τους στόχους μας. Πρέπει όμως να φροντίζουν για επαρκή διαφάνεια, σωστές διαδικασίες, όπως ισχύουν στην εσωτερική αγορά. Οι οδηγίες του 2004 ε, επιτρέπουν να έχουμε αρκετή βεβαιότητα. Συνεπώς, ο Ευρωπαίος νομοθέτης δεν θα πρέπει να νομοθετήσει παρεπτέρω όσον αφορά την Green Public Procurement, GPP. Σίγουρα χρειάζονται εργαλεία, αλλά σίγουρα τα πράσινα κριτήρια πρέπει να έχουν την πρώτη θέση στις δημόσιες συμβάσεις, όπως επίσης και παραδείγματα βέλτιστων ε, πρακτικών που πρέπει να προωθηθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Όμω πρέπει να υπάρχει πιο συστηματικά διαβούλευση με τον κλάδο από ό,τι κατά το παρελθόν. Η νομολογία. Σίγουρα βοηθάει να συμπεριληφθούν και κοινωνικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσει, αρκεί να έχουν άμεση σχέση με το στόχο τη σύμβασή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών που να περιλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις και να μελετήσουμε και την δυνατότητα για ένα νομοθετικό πλαίσιο βάσει αυτής της πρακτικής. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μας οδηγούν σε ένα ερώτημα για το πώς πρέπει να έχουμε νέες ε, προσπάθειες όσον αφορά το in-house procurement, την αυτεπιστασία. Χρειάζεται διευκρίνηση και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διευκρίνηση αυτή. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση. Η Business Europe πιστεύει ότι οι συμβαλόμενες αρχές μπορούν από μόνες τους να προχωρήσουν και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι Δήμοι μπορούν επίσης να οργανώσουν τη συνεργασία όπως εκείνοι θέλουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα τηρούν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρέπει εδώ πέρα να πούμε ότι σύμφωνα με το Δικαστήριο πρέπει να καλύπτονται τρεις προϋποθέσεις, όπως στην περίπτωση Handel. Να υπάρχει συμφέρον προς το κοινό, να μην υπάρχει τρίτη πλευρά και η συνεργασία αυτή να χαρακτηρίζεται από συνεργασία και διάδραση ανάμεσα στους δημόσιους φορούς και να μην είναι ο ένας φορής ο οποίος ε, προσφέρει λύσεις και άλλοι πληρώνουν για αυτή. Για να ολοκληρώσω. Ο ευρωπαϊκό κλάδο πιστεύει ότι δεν πρέπει να ξανανοίξει το θέμα των οδηγιών μόλι πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του. Και όχι επειδή. Δεν είναι επειδή έχουμε κακή νομοθεσία που βλέπουμε κακή εφαρμογή των δημοσίων συμβάσεων. Όχι. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν πολύ σοβαρές παραβιάσεις, αλλά ο λόγος δεν είναι η κακή νομοθεσία, αλλά οι κακές πρακτικές που ισχύουν και η κακή εφαρμογή. Η Business Europe πάντως, εφόσον αποφασιστεί να υπάρξει άνοιγμα των οδηγιών, είναι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Νόστετ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα κάνω την παρουσίασή μου όσον αφορά τη σουηδική εμπειρία. Εργαζόταν με την πράσινη κατοική προμήθεια επί 10 χρόνια Έχω εμπειρία και από άλλα κράτη-μέλη, από την ομάδα του G7, την ομάδα των 7 των πρασίνων, 7 χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή και εργάζονται πάνω στην πράσινη αυτή κρατική προμήθεια και έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έχουμε από το 2003 η Σουηδική κυβέρνηση έχει ένα εργαλείο, δημιουργήσαμε ένα εργαλείο, ένα μέσο για την πράσινη αυτή κρατική προμήθεια στη Σουηδία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ε, κάνει ασχολείται με τον τομέα. Αυτό το μέσο περιέχει σχετικά κριτήρια για διάφορες ομάδες ε, προϊόντων που αγοράζονται συνήθως. Ήταν αρκετά επιτυχής η προσπάθεια. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στον τομέα των κατοικών προμηθειών και τα κριτήρια είναι καλοδιατυπωμένα και ταιριάζουν με τον νόμο περί κρατικών ε, προμηθειών. Επόμενη διαφάνεια. Δεν θεωρούμε ότι η νομοθεσία εν γέννη είναι ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο για να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον στις κρατικές προμήθειες. Όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη διευκρινήσεως, κυρίως αν δείτε τα κοινωνικά κριτήρια και πώς γίνεται η επαλήθευση των ε, κοινωνικών κριτηρίων ειδικά όταν πάμε στα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι πρόβλημα αυτό. Κυρίως τα συστήματα ετικετοθεσίας οικολογικής στις κρατικές προμήθειες είναι πρόβλημα, διότι όλα τα κριτήρια για την οικολογική σήμανση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κρατικές προμήθειες, είναι πολύ περίπλοκα και χρονοβόρα τα συστήματα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει με ένα, μία φωνή οι διάφορες γενικές διευθύνσεις να συντονίζουν τα λεγόμενά τους όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες και βλέπουμε διαφορετικές πρωτοβουλίες από διαφορετικές γενικές α, διευθύνσεις όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις και τις πράσινες κρατικές προμήθειες. Τα κριτήρια για τις ίδιες ομάδες προϊόντων δεν είναι τα ίδια και αυτό είναι απογοητευτικό να το βλέπει κανείς. Βλέπουμε υπάρχει η δυνατότητα εναρμονίσεως των απαιτήσεων για τις προμήθειες όπως τα γενικά προϊόντα, τα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας, πληροφορικής. Θα είναι καλύτερο και για τους προμηθευτές, θα επικρατεί μεγαλύτερη διαφάνεια και θα είναι και πιο κάτω αποτελέσματα για την αγορά εάν όλοι χρησιμοποιούν τα ίδια αναρμονισμένα κριτήρια. Θα είναι μεγαλύτερος αντίκτυπος, οι μεγαλύτερες συνέπειες στην αγορά. Θα είναι πιο ξεκάθαρη η κατεύθυνση προς την οποία θέλει κανείς να κινηθεί. Η μεγάλη πρόκληση είναι να εστιαστούμε σε βιώσιμους πόρους. Να πάμε σε βιώσιμους κρατικές προμήθειες, από GPP, από την πράσινες κρατικές προμήθειες, σε sustainable ε, public procurement. Προς το SPP, αυτός είναι ο στόχος. Δεν ξέρω αν βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες αυτή τη διαφάνεια. Υποτίθεται είναι η αλυσίδα της προμήθειας και αν θέλετε να ακολουθήσετε ανάντι όλη τη διαδικασία στο ορυχείο, στο δάσος που μεγάλωνε το δέντρο υπάρχει πρόβλημα διότι οι πληροφορίες δεν ρέουν η αλυσίδα ιδιοκτησίας αν θέλετε δεν υπάρχει για πολλά προϊόντα, για πολλές πρωτεσίλε. για τα δασοκομικά είναι απλά τα πράγματα διότι υπάρχουν συστήματα πιστοποίηση. για άλλα όμω υλικά όπω είναι τα μέταλλα, το αλουμίνιο άλλα υλικά δεν υπάρχουν πληροφορίες κατά, την, κατά μήκος όλης αλυσίδας. Αυτό είναι πρόκληση, διότι πολλές ομάδες προϊόντων εμπεριέχουν πολλά υλικά που έχουν μεγάλες συνέπειες όσον αφορά το περιβάλλον και για να είναι κανείς πράσινος στις προμήθειες αυτές πρέπει να εξετάσει όλη την αλυσίδα μέχρι την πηγή, μέχρι το ορυχείο. Κάπου χάνεται όμως η διασύνδεση, ο κρίκος που συνδέει τις πληροφορίες και θέματα κλίματος. Και εκεί χρειάζεται να δει όλη την αλυσίδα, από πηγή μέχρι προϊόν και αν αυτό δημιουργεί εμπόδια για το εμπόριο. Υπάρχουν πολλά εκκρεμή ερωτήματα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεως ε, και συντονισμού από πλευράς Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Για να συνοψίσω λοιπόν, η νομοθεσία δεν είναι πρόβλημα κατά την άποψή μου. Η πρακτική εφαρμογή είναι το πρόβλημα. Αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο χρειάζονται απλούστερα εργαλεία, περισσότερους πόρους. Πηγαίνετε μέσα στο νέο επίπεδο, είναι ο τίτλος μιας μελέτης. Ε, το βλέπετε στη διαφάνεια, μπορείτε να το βρείτε στην ισοσελίδα μας αυτό. ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Πολύ χρήσιμες, ενδιαφέρουσες ιδέες που εκφράσατε. Παρατηρήσαμε επίσης ότι διαμαρτύρεστε για έλλειψη συντονισμού όσον αφορά τις κατοικές προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές και αυτό θα το συμπεριλάβει στην εκθεσή της η κυρία Ρίουλη, είμαι σίγουρος. Ε, η Πένι Κλάρκ είναι η επόμενη που θα μας μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Πράγματι, ε, καλύτερη αξία για μας δεν σημαίνει το πιο φθηνό, υπάρχει σχέση μεταξύ καλών υπηρεσιών και αγαθών και καλής ποιότητας εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος. Βλέποντας τι έκαναν τα κράτη-μέλη, κυρίως αυτά τα κοινωνικά κριτήρια στις προμήθειες, είναι μακρά ιστορία, κυρίως σε κάποια κράτη-μέλη, ε, βλέπουμε ότι μετά την οδηγία βλέπουμε να πηγαίνουν προς τα πίσω αντί προς τα μπρος. Οι οδηγίες επιτρέπουν τη συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων στις προμήθειες, αλλά τα κείμενα, το ζουμί κυρίω είναι στι συντολογικέ σκέψει και όχι στο διατακτικό του κειμένου. Συμπεραίνω ότι είναι από του λόγου αυτό για τον οποίο δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε όσον αφορά τι κοινωνικέ προμήθειε, λαμβάνοντα υπόψη παραδόση των κρατών μελών. Και πιστεύω ότι όσον αφορά τι πράσινε κρατικέ προμήθειε, ε, εμφανίζονται προβλήματα που αναφέρθηκαν. Ε, και κυρίως ο τρόπος που παρουσιάζεται τα πράγματα πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά κάποιο τρόπο είναι ενδιαφέρον να τεθεί το ερώτημα. Το θέμα της ασφαλείας δικαίου είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως είναι λυπηρό κατά την άποψή μας. Αν θέλουμε να έχουμε πιο κοινωνική Ευρώπη, πιο πράσινη Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε και σαφέστερες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρκετά από τα συνδικάτα μας έλεγαν ότι τα κράτη-μέλη έχουν σαφείς αρμοδιότητες ε, για πολλούς τομείς και θα πρέπει να προστατεύονται, αλλά νομίζω ότι οι οδηγίες περί προμηθειών τελικά είναι αρνητικό παράδειγμα όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν τον κοινωνικό του τομέα εν τη απουσία θετικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αυτό αντικατοπτρίζει τις διάφορες νομικές παραδόσεις των χωρών. Σε κάποιες χώρες δεν αναφέρονται ρητά στον νόμο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σε άλλες χώρες δεν θα ονειρευόσουν ότι θα έπρεπε ο νόμος να λέει ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα για να γίνουν αυτά. Άρα ήρθε η ώρα οι κοινωνικές προμήθειες να προχωρήσουν. Συμφωνούμε με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρωί για τις νέες αρχές της συνθήκης και για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Είναι αλλαγή η συνθήκη της Αβώνας. Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιοι προσλαλήσαντες δεν το ανέφεραν αυτό στις παρουσιάσεις τους και αυτό δείχνει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν το ότι οι δημόσιες αρχές, τα συνδικάτα, οι εργοδότες όλοι γνωρίζουν τις πιο θετικές πτυχές που απορρέουν από τη συνθήκη της πέρα από τη θετική νομολογία, βλέποντας την ιστοσελίδα τη Γενική Διευθύνσεω Εσωτερική Αγορά και τι ερωτήσει και απαντήσει για τι προμήθειε, δεν βλέπει κανεί τι νέε θετικέ τάσει να αντικατοπτρίζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο το κενό. Ήδη το πρωί αναφέρθηκε η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κοινωνικά κριτήρια ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και εμείς και οι οικονομικές επιδόσεις νομίζουμε ότι είναι κάτι σχετικά εύκολο να εξακριβωθεί. Αν δείτε το ιστορικό ότι αρκετέ από τι υποθέσει στι οποίε βασίστηκε η οικονομική επίδοση έχουν αμφισβητηθεί. Η κοινωνική επίδοση μη θεωρούμε ότι είναι πάντα αφηρημένη και η οικονομική επίδοση είναι πάντα συγκεκριμένη. Τούτου λεχθέντω αρκετοί κοινωνικοί εταίροι στην κλωστή φαντουργία, στο catering, στην θέματα ασφάλεια και στις σχέσεις μας με την τοπική αυτοδίκηση στον κοινωνικό διάλογο, όλοι αυτοί αναφέρθηκαν σε αυτά τα θέματα όσον αφορά την κοινωνική κρατική προμήθεια, έχουν εκπονήσει οδηγούς, έχουν προβεί σε δηλώσεις, έχουν δώσει παραδείγματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν για να διευκρινιστεί τι είναι, ποια είναι τα κοινωνικά κριτήρια, τι είναι οι κοινωνικές κρατικές προμήθειες. Ακόμα περιμένουμε μετά τις οδηγίες για έναν οδηγό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήταν θετική προσθήκη και υποστήριξη αν υπήρχε Τώρα να ε, έθετα κάποια παραδείγματα για τα κοινωνικά κριτήρια θα ήταν χρήσιμο. Θα ανέφερα πρωτίστως την ισότητα των φύλων. Είναι πολύ ισχυρή παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Business Europe, στην ETUC υπάρχουν στα διάφορα κείμενα αναφορές στα σωστά ε, πλαίσια και στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για την ισότητα των φύλων, κοινωνική συνοχή και πάμε στους προστατευμένους χώρους εργασίας, συμφωνίες ένταξης με τους κοινωνικούς εταίρους και συμπερίληψης, ε, δίκαιες αμοιβέ, ισότιμες αμοιβέ. Όλοι αυτοί είναι τομεί, δίκαιη αμοιβή και όλα αυτά, συλλογικές συμβάσεις, Τέλος, η διαφάνεια εξίσου σημαντική δεν είναι μόνο κριτήριο οικονομικό αλλά και κοινωνικό Κατά κάποια έννοια χρειάζεται διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις, τις διαδικασίες, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δίδονται σωστές πληροφορίες και συμμετέχουν επαρκώς οι πολίτες και καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Και τέλος, Πρόεδρε, εδώ προφανώς εξετάζουμε τη διαδικασία της προμήθειας, αλλά σύμφωνα και με όσα είπε η Τροπή Ευρωπαϊκή το πρωί, είμαστε σε μια νέα κατάσταση όσον αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίζει ένα θετικότερο πλαίσιο για τι δημόσιε υπηρεσίε. Θα πρέπει να μα ενδιαφέρουν οι στόχοι και τα αποτελέσματα περισσότερε διαδικασίε και οι συμβάσει παραχωρήσεων καλό παράδειγμα. Το πρωί αναφερθήκαμε στην ασφάλεια δικαίου, αναφερθήκαμε στι διαδικασίε, διερωτηθήκαμε αν ε, αυτές οι παραχωρήσεις δίνουν κάποια αξία προστιθέμενη, ε, εξυπηρετούν τους πολίτες, παρέχουν θέσεις απασχόλησης, πρέπει να καλυφθούν ιδιαίτερα προβλήματα. εσφάλεια δικαίου είναι ένα πράγμα, αλλά αν ακολουθήσουμε προσέγγιση επιλύσεις προβλήματος, πώς προωθούμε τις δημόσιες υπηρεσίες και ποιος είναι ο ρόλος των προμηθειών και ποιος είναι ο ρόλος άλλων διαδικασιών για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, Αυτά νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία αναφέρθηκαν το πρωί στην ακρόαση. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή τους. Uh, Και τέλος, ε, ε, νομίζω ότι έχετε κάποιες διαφάνειες. Ναι, ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ. Πραγματικά, εμείς εκπροσωπούμε την ΣΕΚΟΣ Γιουρού που είναι ένας οργανισμός που εκμετρεύεται 25.000 ε, κατοικίες στην Ευρώπη, 12 με 15% ουσιαστικά. Ακριβώς ε, επειδή μια κατοικία είναι ένα συγκεκριμένο, ένας συγκεκριμένος χώρος, εμείς έχουμε να κάνουμε με τις ε, οδηγίες για τις οποίες συζητάμε σήμερα. Τέσσερα πράγματα Πρώτα απ' όλα, δεν θα σας καθυστερήσω με το χρόνο, τα βλέπετε εδώ. Πάντως αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πάνω απ' όλα να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. και να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες και τα έργα. Έχουμε την κοινωνική κατοικία που καταλαβαίνετε ότι τα κοινωνικά κριτήρια είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την περίπτωση. Από την άλλη μεριά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και ο ορισμός που πρέπει να είναι ευραίος όσον αφορά τις ε, συμβάσεις. Και πρέπει να συνδυάζεται με το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί η σύμβαση. Τώρα, οι κανόνες για τις συμβάσεις παραχώρησης θα μπορούσαν να βοηθήσει κάτι τέτοιο, ένας ε, ορισμός, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε την αίσθηση ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μάλλον η συμφωνία μεταξύ συμβαλόμενων μερών βοηθάει περισσότερο προς το παρόν. Είναι μια δύσκολη υπόθεση πάντως. Το θέμα τώρα της ε, εταιρικής ε, σχέσης, της σύμπραξης οι κατοικίες εξορισμού δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το θέμα της σύμπραξης. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει διάκριση στις προσφορές. Οι συμφωνίες πρέπει καλύτερα να γίνονται αμοιβαία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Και να υπάρχει βέβαια πάντα συνεργασία γιατί είναι μια προστιθέμενη αξία αυτή. Γι' αυτό χρειάζεται σχέση με τις δημοσίες αρχές ή με άλλους οργανισμούς. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν ασχολούμαστε με τις κατοικίες πρέπει να αναλαμβάνονται κάθε τόσο πρωτοβουλίες για αλλαγές, να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Είναι μια συνεχής διαδικασία δηλαδή. Και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Σίγουρα οι βέλτιστες πρακτικές βοηθούν εδώ. Κάτι άλλο έχει να κάνει με το βιώσιμο του έργου. Αυτός ο οποίος επενδύει είναι διαφορετικός από εκείνον ο οποίος τελικά επωφελείται. Δεν είναι απαραίτητα η σχέση μονόδρομη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πλευρά θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει κάτι για να λύνονται τα προβλήματα. Ένα άλλο σημείο έχει να κάνει με την ανάπτυξη στις πόλεις. Η οικοδόμηση κατοικιών συνδέεται άμεσα βέβαια με την ανάπτυξη του χώρου των πόλεων. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι μια σύμβαση βέβαια έργου και είπαμε ότι προκρίνεται το 25%. Σίγουρα η χαμηλότερη τιμή είναι εκείνη που επιλέγεται για να αναπτυχθεί το έργο. Συχνά όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι συνέπειες είναι ότι καταλήγει να υπάρχει μια σχέση με τους πελάτες από την οποία πλήγεται η ποιότητα τελικά, η οποία ποιότητα των κατοικιών είναι πολύ χαμηλότερη από αυτήν που θα επιθυμούσαμε. Σίγουρα είναι ένα έργο που παίρνει πολύ χρόνο. Τα κοινωνικά κριτήρια τώρα. Θα τα περάσω γιατί έχουμε ακούσει πολλά μέχρι τώρα για αυτά, αλλά σίγουρα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά περνάω στα συμπεράσματά μου ευθύ αμέσω, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό ακόμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι κοινωνικές κατοικίες είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Δεν πρόκειται μόνο για ένα εμπορικό στόχο, Πρόκειται και για προσφορά βέβαια εργασίας. Μιλάμε τώρα για έργο το οποίο κρατάει πολλές φορές 10 χρόνια. Η κοινωνική συνοχή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις κατοικίες. Και σίγουρα δεν είναι εύκολο σε μια δημόσια σύμβαση να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Έπειτα είναι το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ εκείνων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Χρειάζεται εδώ πέρα περισσότερη συνεργασία όμως για να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος για όλες τις ε, εμπλεκόμενες πλευρές. Η βιωσιμότητα του έργου είναι κάτι που επίσης έχει μεγάλη σημασία. Οπότε και εδώ θα σταματήσω, Πρόεδρε. Αν δούμε την εμπειρία που έχουμε από τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στις κοινωνικές κατοικίες, οι κατοικίες βρίσκονται σε ευάλωτε περιοχές και γειτονιές. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρόκειται για το συμφέρον της κοινωνίας, είναι στον πυρήνα της υπόθεσης. Ε, και το λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. και να ευχαριστήσω και την κυρία Κλάρκ που μα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο το οποίο ε, μπορείτε να πείτε στου φακέλου σα. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσει. Ε, θα ήθελα να δώσω πέντε λεπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανοίγει ο κατάλογο των ομιλητών. Έχω την κυρία Βερνιό, την κυρία Γκέπχαρτ, τον κύριο Έγγελ. Υπάρχει άλλο από του συναδέλφου που θέλει το λόγο. Υποθέτω ότι η κυρία Ρούλε θα ε, παρέμβει επίση. Ο κύριος Χάνσλικ η κυρία Χάνσλικ θα πάρει το λόγο λίγο αργότερα και η κυρία Βάιλερ. Υπάρχει άλλος? και η κυρία Βάιλερ. Η κυρία Βερνιό, Γκέπχαρτ, Έγκλ, Βάιλερ, Ρούιλερ. Η κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ και που προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Εννοείται ότι όταν προσπαθεί κάποιος να απαντήσει σε ερωτήσεις, δημιουργεί και άλλες. Η συνάντηση αυτή μου θυμίζει πολλές συναντήσεις που είχαμε στο παρελθόν και εδώ κοιτάζω την κυρία Γκέπαρτ, γιατί <clears throat> είχαμε δύο τρόπους σκέψης. Από τη μια μεριά είχαμε τους εμπειρογνώμονες που λέγανε ότι υπάρχουσες οδηγίες ε, δεν είναι και άσχημες, δεν χρειάζεται παρετέρω ρύθμιση. Απλώς χρειάζεται βελτίωση στην πράξη, στην πρακτική. Και από την άλλη έχουμε εμπειρογνώμονες, και εδώ έχω στο κατω μια άποψη, έτσι. Εκτίμησα και την κυρία Κλάκ και τον κύριο Δικιόγκ και τον κύριο Ροντρίκης, που λένε έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, τη θελήσαμε και την έχουμε, έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, ακριβώς ώστε η Ευρώπη να είναι πιο κοινωνική και να μπορεί να προστατεύσει περισσότερο το περιβάλλον. Και όταν μιλάω για περιβάλλον, ενώ και το φυσικό χώρο μέσα στον οποίο ζούμε, αλλά και το κοινωνικό μας περίγυρο. <clears throat> Οι κακές πρακτικές υπάρχουν. Έχουμε συνεργαστεί και παρόλα αυτά δεν έχουν λυθεί οι κακές πρακτικές. Όταν ε, είχαμε τις δημόσιες συμβάσεις, κάποια στιγμή εγώ ήμουν αναπληρώτα για θέματα σχολείων, ε, γεμάτο κτλ. Όταν εγώ αποφάσισα για το καλύτερο, γιατί υπήρχαν και κοινωνικά κριτήρια, απασχόληση για παράδειγμα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει κτλ. τα στην περιοχή μου, έπρεπε να το αιτιολογήσω με χίλιου δυο τρόπου. Λοιπόν, τα μέσα που μα δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά να έχουμε μια μέθοδο για να ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Πριν ακούσαμε για την διάρθρωση με τις εξελίξεις και την πρακτική. Εγώ δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν να αποφύγουμε ένα κείμενο το οποίο πολύ συγκεκριμένα να μας λέει περί τίνος πρόκειται και να μας βοηθάει. Μιλάμε εδώ πέρα για θεμητό ανταγωνισμό, όχι για αθέμητο. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται διευκρίνηση για να έχουμε και νομική βεβαιότητα, τόσο οι πολίτες, όσο και επιχειρήσεις, αλλά και οι δήμοι ένα νέο κείμενο που να διευκρινίζει ξεκάθαρα τα πράγματα βάσει της εθήκης της Λισαβόνας και που να μας δίνει και τον τρόπο λειτουργίας θα βοηθούσε. Εγώ ως νομοθέτης δεν είμαι ικανοποιημένη με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δηλαδή δεν μου φτάνουν για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ευχαριστούμε κύριε Γκέπαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορώ να ε, συνεχίσω πολύ ομαλά την παρέμβαση αυτή. Στις τέσσερις παρεμβάσεις που μόλις ακούσαμε, δύο πτυχές τονίστηκαν ιδιαίτερα κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, το πεδίο εφαρμογής των ε, οδηγιών ε, για τις δημόσιες συμβάσεις και η συνθήκη της Λισαβόνας που μας δίνει νέους ε, τρόπους ε, για να ε, διαχειριστούμε, για παράδειγμα, τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε με συνέπεια τις προεκτάσεις του θέματος αυτού. Το δεύτερο θέμα είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την ανάθεση συμβάσεων, ιδιαίτερα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια συμμετείχα στην εισαγωγή των κριτηρίων αυτών στο δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων τότε που είχαμε πολύ έντονε συζητήσει σχετικά με το αν χρειαζόμαστε τέτοια κριτήρια και εάν ναι, εάν θα πρέπει να είναι προαιρετικά ή δεσμευτικά. ως σοσιαλδημοκράτησα αλλά και ως Γερμανίδα ευρωβουλευτής ε, ήμουνα σε διχασμό διότι η, ε, η σοσιαλδημοκράτρια μέσα μου λέει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα κριτήρια αυτά. Η Γερμανίδα μέσα μου έλεγε ότι έχουμε την ε, τοπική αυτοδιοίκηση και θα πρέπει οι Δήμοι μόνοι τους να αποφασίζουν τι θέλουν. βέβαια τελικά η δεύτερη πτυχή κέρδισε και αυτό το βρίσκω σωστό. Ωστόσο, ξεκίνησαν τα προβλήματα κατά την εφαρμογή πώ αποφασίζονται, πώ ορίζονται τα κριτήρια αυτά και αυτή είναι μια συμπληρωματική ερώτηση προ όλου του ομιλητές και πώς μπορούμε παρόλα αυτά να φροντίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει συνοχή ακόμα και αν δεν ορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κριτήρια αυτά και αφήσουμε το θέμα αυτό ε, τελείως στις ε, δημοτικές αυτοδιοικήσεις. Πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό. Κύριο Σέγγελ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή όσον αφορά την τοπική αυτονομία και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι είναι καλό που παγιώνεται για πολλωστή φορά. Αυτό που κάνει είναι ότι παγιώνει όμως τις τοπικές ανεπάρκειες. Είναι αποδεδειγμένο ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στις περισσότερες χώρες οι κοινότητες είναι τόσο μικρές που είναι αδύνατον να επομιστούν τις πιο βασικές αρμοδιότητες και η διακοινωτική συνεργασία ε, δεν είναι τόσο εφικτή γιατί έχουν γίνει πολύ μικρές οι κοινότητες για τις φιλοδοξίες της. Είναι κάτι που δεν άπτεται της εσωτερικής αγοράς αλλά χρειάστηκα, κανένα για να το πω. Είναι συμβάσεις οι δημόσιες ε, προμήθειες και εφόσον είναι συμβάσεις βασική μέρημνα θεωρώ ότι είναι να επικρατεί ασφάλεια δικαίου και όπως αποδεικνύει η ακρόαση και άλλα στοιχεία πριν από αυτό, δεν είναι κάτι, δεν αρκεί αυτή η ασφάλεια που παρέχεται για την ώρα. Για να αυξηθεί η ασφάλεια χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία. Εκεί δεν έχουμε δεσπίσει νομοθεσία ακόμα, στα κομμάτια που δεν έχουμε νομοθετήσει. Επιβεώνεται το γνωστό δίλημα. Αντίθεση αύξηση ασφαλεία δικαίου μέσω περισσότερη δεσμευτική νομοθεσία ή να μην αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου. Και αυτό που δεν ρυθμίζεται μέσω συμβάσεως και μέσω του νομικού πλαισίου ε, οδηγεί στο δικαστήριο. Δηλαδή είναι ο πολιτισμός της αμφισβήτητης και της προσφυγής. Νομίζω ότι δεν θα ξεφύγουμε από αυτό ούτε στο μέλλον. Προσωπικό συμπέρασμα ήταν από αυτά που άκουσα σήμερα, περισσότερο παλά ερώτημα. Κάθε ερώτηση οδηγεί σε αντιφατικές απαντήσεις, πιστεύω, σχετικά με αυτά που έλεγα, οπότε δεν θα θέσω ερωτήσεις για να μην δημιουργήσω νέες αντιφάσεις μέσα των απαντήσεων. Η ε, κυρία Βάιλερ. Πολύ σωστά υπόθηκε αυτό, αν μεταφράστηκε σωστά. Ε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ε, κουλτούρα των διαμαχών, ε, ούτε πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι αποτελεί ε, ένα από τα στηρίγματα της ε, δημοκρατίας. Η κυρία Κέπχαρτ μίλησε για διχασμό ε, και εγώ ως πρώην δημοτική πολιτικός πιστεύω ότι θα πρέπει πράγματι οι δήμοι να αποφασίζουν. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ε, δημοτικές αρχές εφόσον έχουν, τις αρκεί, τις, ε, εφόσον έχουν ε, επαρκείς γνώσεις. Αλλά Πολλοί, δήμοι δεν τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν 13 ε, κριτήρια. Αναφέρθηκαν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Και οι γνώσει αυτέ είναι απαραίτητε για να αποφασίσουν οι δημοτικοί πολιτικοί ποια κριτήρια θέλουν να εφαρμόσουν. Δεν χρειάζεται να εφαρμόσουν όλα μαζί. Ε, θα πρέπει να θέσουν προτεραιότητε. Και πιστεύω δεν έχουμε κάνει ψηφοφορία, αλλά ομολογώ ότι δεν θέλω ε, δεσμευτική και απόφαση του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της επικουρικότητας. Μπορεί οι συνάδελφοί μας στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος λόγω του θέματος του κλίματος σε τρία-τέσσερα χρόνια να ε, εφαρμόσουν υποχρεωτικά τα κριτήρια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό και ούτε θα ήθελα να θέσω τέτοια πρωτοβουλία. Ωστόσο, επειδή διαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων, έλλειψη πληροφόρησης, θα ήθελα να αναφερθώ στο παράδειγμα παράδειγμα των Σουηδών που είπαν ότι έχουν εκπονήσει κατευθυντήριε γραμμέ, βέλτιστε πρακτικέ και νομίζω ότι έχουν προχωρήσει πολύ πιο πέρα από όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Ε, ίσως θα ήταν οι εμπειρίε του χρήσιμε για τι κατευθυντήριε γραμμέ. Κατευθυντήριε γραμμέ όμω, όχι ε, νομοθεσία από την Κομισιόν για να, ε, για να διαδοθεί καλύτερα η γνώση σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Οι δήμοι οι άνθρωποι λένε ότι αν ο Δήμο θέλει να προωθήσει, για παράδειγμα, τις ε, γυναίκες, ε, τότε θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος ο Δήμο. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσουν οι πολιτικοί ε, των Δήμων. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρούλε και μετά να ακούσουμε τους, ε, τους ομιλητές μας. Ήθελα να εξοικονομήσω λίγο χρόνο και γι' αυτό ε, ε, θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις και προς την Κομισιόν. Ε, ωστόσο, ε, θέτω ερωτήσεις και προς τους συμμετέχοντες αυτού του κύκλου. Ε, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει ε, επαρκής ε, συντονισμός εντός της Κομισιόν, δεν υπάρχει καλή πολιτική πληροφόρηση και δεν υπάρχει σωστή κατανόηση. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πληροφορίες για όλα τα κριτήρια σε μία ιστοσελίδα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, στις ε, τοπικές αρχές για να, ενισχύσουμε, για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη διαδικασία. Μία ερώτηση προς την Νορβηγίδα ε, ομιλήτρια. Έχω την εντύπωση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν από το καθεστώς, έχουν παραπονεθεί σε μένα λόγω του υψηλού κόστους, λένε ότι είναι υπερβολικά πολύπλοκες οι διαδικασίες, ότι χρειάζονται ε, ακριβή νομική συμβουλή ε, εξωτερική κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Ε, θα σας δώσουμε και λίγο χρόνο να σκεφτείτε και μετά θα δώσω το λόγο το πολύ για πέντε λεπτά στον ε, κύριο Βίτνερ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε και περαιτέρω δυνατότητες ανταλλαγής, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τη θέση σας κατόπιν η κυρία Χάνσλικ και η κυρία Ρούλε που θα συνοψίσει τη συζήτηση. Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα αυτά μέχρι τις 12.30. Ναι. Η κυρία Τζίνες πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ε, ξεκινήσω με την ερώτηση της κυρίας Ριούλε που σχετίζεται με την, το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, στη Νορβηγία εκπονήσαμε μελέτη ε, όπου εξετάζεται το διοικητικό άχθος και η ανταγωνιστικότητα και Καταλήξαμε ε, στο ποσό 60.000 ευρώ, δηλαδή στην ε, Νορβηγία το κατόφλι για ε, την συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις είναι 60.000 ευρώ. Και αυτό με οδηγεί στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αγορά. Και ξέρω ότι είναι καυτό το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκές χώρες επίσης. Αλλά ας εξετάσουμε τις σκανδιναβικές χώρες. Η Δανία έχει το ίδιο κατόφλι με την Ορβηγία. Η Σουηδία σκοπεύει να ε, εισάγει ακόμα χαμηλότερο κατόφλι αν περάσει από το Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουν οι ευρωβουλευτές. Εάν θέλετε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις, ε, προσφορές για ε, δημόσιες συμβάσεις, μην κλείνετε την αγορά, αλλά θα πρέπει να ξέρουν πού θα βρουν τις σχετικές πληροφορίες. Η δημοσίευση είναι η λέξη κλειδί. Επόμενη ερώτηση που θα θέλω να απαντήσω, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την συνέπεια. Κατευθυντήριε γραμμέ, εξηγήσει, παραδείγματα, ένα βιβλίο μαγειρική σαν να λέμε. Και τελικά θα πρέπει οι αναθέτουσε αρχές να, απο... να διαλέξουν τι συνταγέ που θα μπουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούιλε νομίζω ότι σύντομα θα συγγράψει αυτό το βιβλίο μαγειρική. Ο κύριο Νόστετ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναπτύξω το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα φιλόδοξα περιβαλλοντικά κριτήρια αποτελούν εμπόδιο. Μάλλον ρωτήσαμε αν είναι, ε, ε, αν είναι εμπόδιο και είπαν ότι όχι. Ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν επικεντρώνονται οι αρχές στην τιμή. Ως πρόεδρος της άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής της Κομισιόν, όπου συμμετέχουν 7 χώρες, που θα βοηθήσει την Επιτροπή στις εργασίες ε, για τις συμπράξεις δημοσίου δικαίου. Ε, ε, πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για μια βιώσιμη πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβόσεων. κυρία Κλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κερδίσω τις συνθήκες αγώνας. Ναι, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχεται Τώρα, τι ουσίες θα χρησιμοποιήσουμε για το τζελεμεντέ μας. Ε, έχουμε συζητήσει με πράσινες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, κοινωνικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε όλους αυτούς. Υπάρχουν αποστάσεις όμως μεταξύ του εθελοντικού και του υποχρεωτικού. Το θα έπρεπε, τους στόχους, βέλτιστη πρακτική, στόχους και οι στόχοι είναι κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και πρόοδος στους αλλά είναι η έλλειψη συνέπειας δεν είναι το πρόβλημα. Και η Νορβηγία συζητά και την ε, διάσκεψη, ε, τη σύμβαση του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που είναι υποχρεωτικό αντισβεστικό. και πολλα κάτι κράτη-μέλη έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση και νομίζω ότι είναι κάτι που θα εφαρμοστεί και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, διαφορετικά πράγματα και με τα χαράς να επεξεργαστούμε περαιτέρω το θέμα, όπω έκανε και το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν, και να συνεχιστούν και συζητήσει. Δεν θα πρέπει να λέμε ότι ε, επί το ότι δεν έχουμε προχωρήσει σήμερα πιο πολύ από ό,τι έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, είναι λανθασμένη ανταπόκριση της όλης δουλειάς που έχουμε γίνει. Έχουμε εντολή που μας δόθηκε, έχουμε κάποια μέσα, απλώς δεν έχουμε οικοδομήσει επαρκώς. Κύριος Διόμ. Δύο μικρές παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτα απ' όλα για τη διευκρίνηση της ρύθμισης, περισσότερη ρύθμιση, συντονισμός κτλ. Βέβαια, πολλά είπατε για αυτά. Βοηθάνε, αλλά δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα. Και το βασικό πρόβλημα, προσπάθησα να σας εξηγήσω, είναι ότι οι κανόνες των δημοσίων συμβάσεων δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στα μέρη που συμμετέχουν, ενώ χρειάζεται συνοχή Πρέπει όλοι να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, σε ένα ίδιο project. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Οπότε γι' αυτό μίλησα για ισορροπία. Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ουσιαστικές στις γειτονιές. Πρέπει να συμμετέχουν για να δημιουργείται η κοινωνική συνοχή στις γειτονιές. Βγαίνουν όμως από το σύστημα, το ακούσαμε και εδώ. Βλέπουμε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Ενώ θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υιοθετούνται μέτρα που να βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις στις γειτονιές τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ λοιπόν και αυτό το πάνελ για τα τόσα χρήσιμα και ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ελπίζω να συνεχίσετε τη δουλειά σας σε αυτό το θέμα και θέλω να πω σε όλους σας ότι η συνεισφορά σας μας βοηθάει να κατανοούμε από τη μια καλύτερα τα όσα εξετάζουμε, από την άλλη βέβαια μας δημιουργούν και νέες απορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά και με την Επιτροπή και εδώ μιλάω εκ μέρους νομίζω όλων των πολιτικών ομάδων, αυτό που μας ενδιαφέρει στην Επιτροπή μας είναι να πάμε μπροστά, να προχωρήσουμε. Και ακόμα κι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας επιτρέπει να έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν ξέρω ο κύριος Βίκμαν αν θα μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τέλο πάντων, θα του δώσω τρία λεπτά για να μας πείτε για αυτά που ακούσατε, ξέρετε ότι δεν θα τα καλύψετε όλα. Είναι πάντα ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρίσκεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα για μας. Κάτι που πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή είναι ότι, όπω είπατε και πριν, περιμένουμε την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, ό,τι και να πω εγώ τώρα, καταλαβαίνετε, θα εξαρτηθεί από τη συνέχεια, από την ε, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σρόσκα θα μοιραστεί την παρέμβαση της Κομισιόν σήμερα, οπότε ξεκινάω εγώ. Και ξεκινάμε το δεύτερο γύρο για το θέμα των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι αλήθεια ότι είχαμε πολλές πρωτοβουλίες από διάφορες πλευρές, ιδιαίτερα όσον αφορά το μη υποχρεωτικό δίκαιο, το soft law. Υπάρχει βεβαιότητα, ακούσαμε. Δυσκολίες στις δημόσιες αρχές, ακόμα και για πρόσβαση έγγραφα πολλές φορές. Εμείς δουλεύουμε και το πρώτο που θα φροντίσουμε για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανακοίνωση η οποία θα συγκεντρώνει όλα αυτά τα πράγματα ώστε οι αρχές να καταλαβαίνουν πιο εύκολα τι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εφαρμόζουν, ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθούν εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κάποια δημόσια σύμβαση. Αυτό θα φροντίσουμε να το συγκεντρώσουμε και θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε με τη νέα θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχρόνως, θα έχουμε και τομιακές κατευθυντήριες γραμμές για τα κοινωνικά, για παράδειγμα, σύντομα μάλιστα. Και θα είναι πιο πρακτικός οδηγός. Θα δείχνει σε ποιο στάδιο της διαδικασίας μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κοινωνικά κριτήρια και πώς οι εντάσεις που έχουμε συνήθως είναι ότι από τη μια μεριά θέλουμε ε, θεμητές ε, δίκες ε, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες και από την άλλη μεριά θέλουμε συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων. Θα φροντίσουμε λοιπόν για την πρακτική εφαρμογή, το στάδιο της πρακτικής εφαρμογής. Κάτι άλλο σύντομα για εργαστήρια και την εθελοντική βάση. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει στην οδηγία, ότι καλύπτεται και ότι μπορούμε να ευνοήσουμε τη δημιουργία και την εργα... τη δουλειά τέτοιων ε, εργαστηρίων. Γενικότερα τώρα για το ότι υπάρχουν ε, υπερβολικά πολλοί κανόνες και είναι πολύ περίπλοκοι. Θέλουμε από τη μια ε, ευελιξία και από την άλλη διαφάνεια η εσωτερική αγορά. Για να δουλέψει όμως χρειάζεται κάποιους κανόνες που να είναι ίδιοι για όλους. Για να ξέρουν όλοι πώς μπορούν να συμμετέχουν με εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη μία χώρα σε κάποια άλλη χώρα. Σήμερα ακούσαμε ότι για άλλους είναι αυστηροί οι κανόνες, για άλλους δεν είναι αρκετοί. Γι' αυτό και μιλάμε για ισορροπία. Χρειάζεται η σωστή ισορροπία. Κάποιοι πάντως από αυτούς τους κανόνες έχουν να κάνουν με το εθνικό δίκαιο Ακούσαμε πολλά πράγματα και για το εθνικό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε ε, να θαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Τέλος, η αίτηση για μια τέλος ενδιαφέροντος για μια ε, δημόσια σύμβαση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι η κατάρτιση βοηθάει πάρα πολύ για να γίνεται αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Θα προσπαθήσω να τονίσω κάποια από τα σημαντικότερα σημεία όσον αφορά τις συμβάσεις παραχωρήσεων και τις, ε, ε, τη συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα και θα πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερέστερα συγκεκριμένα ζητήματα υπό η αδίποτε ενδεδειγμένη μορφή. Βεβαίως γνωρίζετε πολύ καλά όλα τα προβλήματα και όλες τις ανησυχίες που εθίγησαν άλλο στη σημερινή συζήτηση. Και αυτό είναι κάτι που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι περαιτέρω προβληματισμό σίγουρα απαιτείται πρέπει να δούμε πώς θα επιφέρουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον τομέα. Και συζήτηση για τις συμβάσει παραχωρήσεων δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκίνησε προετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξεπώνησε δύο ανακοινώσει. Είχαμε και από πλευρά Κοινοβουλίου συνεισφορά με την έκθεσή του του 2006 που το Κοινοβούλιο εξέφρασε ενδιαφέρον για νομοθετικά μέτρα στον τομέα. Πολλή δουλειά έχει γίνει. Βεβαίω θα πρέπει να συνεχιστεί. διερωτώμεθα τα ίδια ερωτήματα, όπως και εσείς. Γιατί συμβάσει παραχωρήσεων που είναι κάτι περιπλοκότατο, με μεγάλη προστιθέμενη αξία και που ήταν επανειλημμένα αντικείμενο της νομολογίας του δικαστηρίου, γιατί δεν καλύπτονται πλήρως ή επαρκώς. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε τα αναπομένοντα κενά τα εκκρεμή προβλήματα, οι οδήποτε κανόνες ή οδήποτε μέτρα που θα υιοθετηθούν στο μέλλον, βεβαίως θα πρέπει να περιέχουν απλότητα και ευελιξία. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε το άχθος μέσω νέων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί καθεαυτοί δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την ευελιξία της συμβαλόμενης αρχής. Χρειάζεται σωστή ισορροπία. Πρέπει όμω κάτι να γίνει, αυτό καταλαβαίνουμε. Ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την όλη ανάλυση. Ξεκίνησε η διαδικασία των συζητήσεων και προβληματισμού για το επόμενο βήμα, χωρί να προδικάζουμε το αποτέλεσμα όσον αφορά το περιεχόμενο τη μορφή τη εκθέσεω αξιολογήσεω και πιστεύω ότι θα κάνουμε κάποιε προτάσει στα μέσα του έτου. Όσον αφορά τη συνεργασία δημόσιου-δημοσίου, οι κανόνες των ε, κρατικών συμβάσεων δεν αναμειγνύονται στην ελευθερία των δημοσίων αρχών να στραφούν προς την αγορά όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Υπάρχει ανεξαρτησία όσον αφορά την επιλογή των ε, αρχών των που αναθέτουν το έργο όσον αφορά τις αποφάσεις του δικαστηριού. Ρίχνουν κάποιο φως, υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε. Ξεκινήσαμε συζήτηση με τα κράτη-μέλη για την καλύτερη δυνατή λύση για διευκρίνηση των αποφάσεων που ελήφθησαν για να βρούμε την καλύτερη βιώσιμη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο και τους δύο. Είμαι σίγουρος ότι η δουλειά μας θα συμβάλλει στο διάλογο και θέλουμε να διατηρήσουμε διάλογο με τα κράτη-μέλη και με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Κάτι που κάναμε και χθε πάνω σε άλλο ζήτημα. Οι διερμηνείς μας δίνουν λίγο ακόμα χρόνο και του ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφου να συνοψίσουν σύντομα, ίσως ένα δίλεπτο ο καθένας. Μπορεί έχετε δύο λεπτά, εσείς όλου ιδιαίτερος. Η συγγήτριά μας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, τους φιλοξενούμενους μας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις τους. Όπως είπατε, είμαι σκιώδης συγγήτρια στην Επιτροπή Ίντερ και θα ήθελα να θέσω το θέμα της συνεργασίας με τρίτες χώρες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Θα ήθελα να τονίσω τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εσωτερικής μας αγοράς και των διεθνών αγορών. Νομίζω ότι είναι κάτι προφανές και δεν πρέπει να λησμονείται. Οι δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα το διεθνές δίκαιο, διέπονται από πολυμερείς συμφωνίες. Όχι όμως όλα τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ συμμετέχουν σε αυτές τις πολυμερείς συμφωνίες, μόνο οι ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης, διμερείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες οδηγούν στη σύναψη συμφωνιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Εδώ έχω υπόψη μου τη Χιλή και το Μεξικό. Ποιο είναι το ζουμί ότι με κάποιες εμπορικούς εταίρους δεν έχουμε συμφωνία όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Αυτοί οι εταίροι όμως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουν πρόσβαση στις δικές μας αγορές από τη στιγμή που πληρούνται κάποια κριτήρια βεβαίως. Όμως αυτοί οι εταίροι από την άλλη, από την πλευρά τους εμποδίζουν τη δική μας πρόσβαση στις δικές τους αγορές. Και εδώ αναφέρομαι στην Κίνα. Να τονίσω όμως ότι και εταίροι με τους οποίους έχουμε δεσμευτικές συμφωνίες και αυτοί προσπαθούν να εμποδίσουν τη δική μας πρόσβαση στις δικές τους αγορές όπως είναι ο Καναδάς ή η Ιαπωνία. Λοιπόν, δημόσιες συμβάσεις έχουν μεγάλο δυναμικό για μας, είναι πηγή δυνατοτήτων για μας και ευκαιριών. Οι εταιρείε μας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όμως πλήρως το δυναμικό αυτό και αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Διότι αυτές οι εταιρείε δεν έχουν επαρκές ρευστό να δαπανίσουν ούτως ώστε να τους ανατεθούν δημόσια συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να τηρείται η αρχή της αμοιβαιότητας. Θα έπρεπε να περιορίσουμε την πρόσβαση στις δικές μας αγορές δημοσίων συμβάσεων σε εκείνους τους εταίρους από τρίτες χώρες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές μας αγορές αλλά δεν μας δίνουν πρόσβαση στις δικές τους αγορές. Τι ούτω τρόπος πιστεύω ότι θα τους δώσουμε κάποια κίνητρα ούτω ώστε να ανοίξουν την αγορά τους των δημοσίων συμβάσεων στις δικές μας εταιρείες. Πρέπει να γίνουν πολλά για να χρησιμοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αυτό και εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε διεθνές επίπεδο. Φοβούμε ότι οι εταίροι μας στον κόσμο δεν μοιράζονται εν γέννη την πεποίθησή μου. Οι περισσότεροι εταίροι μας εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση τη δική μα στις δικές τους αγορές. Ευχαριστώ που μας δώσατε μια πρώτη γεύση όσον αφορά την πληρέστατη γνωμοδότησή σας. Η Χάιντι Ρούλε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, πολύ και να ε, συμφωνήσω με αυτό που είπε η Σίτρια ότι πολύ συχνά σε τέτοιες ε, ακροάσεις πιο πολλές ερωτήσεις τίθενται παρά απαντήσεις. Τέσσερις σελίδες ε, κείμενο έχω, οι αιτιολογικές σκέψεις ε, πιάνουν ήδη μία σελίδα. Δύο μισή σελίδες ουσιαστικά είναι το ζουμί του, της έκθεσης. Ε, σας το λέω για να μην έχετε υπερβολικές προσδοκίες από την έκθεσή μου, διότι ναι, σίγουρα θα άξιζε τον κόπο να γράψουμε μαγείο, βιβλίο μαγειρική, συγγνώμη, αλλά σίγουρα δεν αρκούν τέσσερις σελίδες για κάτι τέτοιο. Ε, εγώ θα ήθελα να κλείσω την ακρόαση ευχαριστώντας ε, Χάιντι που ηγήθηκε στις διαδικασίες αυτής ε, και που ήσουν τόσο ανοιχτή απέναντι σε όλους. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να επιφέρουμε πολύ θεμένη αξία. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν και λυπάμαι που δεν είχαμε την αίθουσα που έχουμε συνήθω. Ε, μην σα πω κιόλα ότι ε, κάνει κρύο σε αυτή τη μεριά τη αίθουσα. Η Επιτροπή μα θα ξανασυναντηθεί το απόγευμα σε άλλη ε, αίθουσα συνεδρίαση που ελπίζω θα είναι πιο ζεστή, στην 3C050. Η ωραία τούτη εδώ μικρή αίθουσα λοιπόν θα αντικατασταθεί από μια μεγάλη και θα είναι ο Γενικό Γραμματέα τη Ισπανία για την πολιτική καταναλωτών θα τα πούμε στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ πολύ.